Καλημέρα σας. Καλημέρα αυτοί που έχουν έρθει στην ώρα τους δεν πρέπει να υποστούν κυρώσεις για την ευσυνειδησία τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. So, wir hatten gestern ja keinen Koordinator. Δεν κάναμε συνεδρίαση των συντονιστών όπως ξέρετε, επομένω δεν μπορώ να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης. Είπαμε ότι έχει αναβληθεί η συνεδρίαση μέχρι τις 25 Ιανουαρίου των συντονιστών. Aber am 7. Είχαμε όμως μια συνεδρίαση συντονιστών στις 7 Δεκεμβρίου και υπάρχουν τα πρακτικά αν, ε, από αυτή τη συνεδρίαση. Αν έχετε κάποια αντίληση πρέπει να μα το πείτε. Περνάμε στο σημερινό πρώτο σημείο. Έλεγχος εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, παρουσίαση από την DigiMove της εκτελεστικής πράξης για τους κανόνες που αφορούν τη χρήση οπισθίων αεροδυναμικών διατάξεων, τα λεγόμενα οπίστια πτερίγια. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του κειμένου αυτού. Η οδηγία 719 του 2015 που έχουμε μόλις εγκρίνει την Άνοιξη ε, προβλέπει να υπάρχει δυνατότητα οπιστίων πτεργίων στα οπίστια των φορτηγών αυτοκίνητων για να βελτιωθεί η αεροδυναμική τους απόδοση. Το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής λέει ότι πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Καταρχήν, η Move θα πρέπει να εκδώσει μια εκτελεστική πράξη για τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών των κανόνων για τα πτερία και δεύτερον η DG Grow θα πρέπει να αναθεωρήσει τους κανόνες για την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων οχημάτων, ώστε τα προϊόντα αυτά να μπορέσουν να εγκριθούν πριν τεθούν στην αγορά. Σε ό,τι αφορά την δική μας ε, απόφαση, εμείς έχουμε συναθρήσει μια ομάδα από πυρογνώμονες που προέρχονται από όλους τους ε, το εμπλεκόμενους τομείς, κατέληξαν σε μια σειρά συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά την έγκριση των εξαρτημάτων αυτών και τις συνθήκες χρήσης τους. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε σε ορισμένα πορίσματα και η DigiMove έχει <clears throat> συμπεριλά αυτά τα στοιχεία στην εκτελεστική πράξη. Αυτή η εκτελεστική πράξη είναι το αντικείμενο της σημαίνει συζήτησης. Έχει παρουσιαστεί στην Επιτροπή Επιτροπολογίας των Κράτων Μέλων στις 30 Οκτωβρίου και η Επιτροπή Επιτροπολογίας έχει ε, καταθέσει μια πρόταση αναμένοντας την πρόταση της Desert Grow η οποία επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα αυτό με εμπειρογνώμονες σε σχέση με την εκτελεστική αυτή πράξη και υπολογίζει ότι το, την άνοιξη θα έχει τελειώσει την εργασία της. Επομένως προς το τέλος του, της άνοιξης το πολύ πολύ των ε, Ιούνιο θα έχουμε και τις δύο αυτές πράξεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν στην έγκριση των κρατών μελών σε δύο διαφορετικές επιτροπές την Επιτροπή για τα Φορτηγά που αφορά την DigiGrow <coughs> και την Επιτροπή Μεταφορών για την DigiMove. Και μετά <coughs> το, τα δύο αυτά κείμενα θα εγκριθούν ταυτόχρονα προς όφελος των ταλικέριων. Επίσης, Θέλω να σας διευκρινίσω, διότι σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι στο κείμενο της οδηγίας προβλέπεται να υπάρξει μια βελτίωση το εμπροστίου προφίλ των οχημάτων. Και για το θέμα αυτό η DG Grow θα πρέπει να προτείνει <clears throat> μια αναθεώρηση, μια αναδιαμόρφωση όλων των κανόνων που ισχύουν μέχρι στιγμής. Εγώ ήρθα σε επαφή με την DG Grow, η οποία <clears throat> επιβεβαίωσε ότι είχε αναλάβει την ευθύνη κατά τη διάρκεια, <clears throat> όπως έκανε κατά τη διάρκεια του τριλόγου πέρσι, να παρουσιάσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν από το τέλος του 2016 ένα σύνολο στοιχείων σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, ώστε το ταχύτερο δυνατό οι εταιρείε που παράγουν φορτηγά αυτοκίνητα να μπορέσουν να κάνουν τις σχετικές μελέτες και να μπορέσουν να θέσουν στην αγορά τον εξοπλισμό αυτό μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία. Ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάζεται να απαντήσουμε είναι το ερώτημα των λεγόμενων 20 εκατοστών. Ξέρουμε ότι όταν ο εξοπλισμός αυτός των πτερυγίων που τίθενται στο πίσω μέρος των οχημάτων όταν αναδιπλώνονται, έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να ξεπερνούν τα 20 εκατοστά πλέον του μήκους του οχήματος, ώστε να μπορούν να τεθούν σε ε, φαγόνια μέσα στα πλαίσια των συνδυασμένων μεταφορών. Στην εκτελεστική πράξη όμως έχουμε προσθέσει και μία σύντομη φράση που λέει ότι αυτή η προϋπόθεση ισχύει εάν το φορτηγό αυτό όχημα προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό ξέρω ότι θα οδηγήσει σε διαμάχες και θέλω να εξηγήσω γιατί έχουμε προσθέσει μια τέτοια φράση. Μέσα στα πλαίσια της ομάδας εμπειρογνωμόνων υπήρξαν ορισμένοι επιστήμονες και βιομήχανοι ότι είπαν ότι σήμερα όλα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σήμερα στην αγορά όλα τα προϊόντα τα οποία είναι εν εξελίξη θα <clears throat> εκπληρώσουν την προϋπόθεση των 20 εκατοστών. Μπορεί όμως σε 5, 10, 15 χρόνια να υπάρξει εξέλιξη της τεχνολογίας που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία θα είναι πιο αποτελεσματικά από τα τωρινά προϊόντα, τα οποία όμως δεν θα ικανοποιούν την προϋπόθεση των 20 εκατοστών. Θα πρέπει λοιπόν ως εκ τούτου να εμποδίσουμε την πρόοδο της τεχνολογίας για αυτά τα 20 εκατοστά ή θα πρέπει να <clears throat> εξασφαλίσουμε ότι αν κάποιος μεταφορέας θέλει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του σε ένα ε, βαγόνι σιδηροδρομικό να έχει δυνατότητα να αφαιρέσει τον εξοπλισμό αυτό για να μπορεί να χωράει το όχημα του στο βαγόνι. Γι' αυτό έχουμε προσθέσει αυτή τη μικρή φράση. Για μας αυτή η μικρή φράση δεν εμποδίζει τις συνδυασμένε μεταφορές. Ξέρετε πόσο προσφυλή στην Κομισιόν είναι οι συνδυασμένες μεταφορές. Δεν θα υπάρξει λοιπόν κανένα πρόβλημα και αν υπήρχε δεν θα το θέταμε αυτό στο κείμενο. <clears throat> Επίση, ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει μια διαφορετική άποψη και θέλει να εξαφανιστεί αυτό το, ε, το τμήμα της φράση εάν είναι πραγματι έτσι θα εξαφανιστεί. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κανένα σχόλιο από τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν μπορώ να σας πω προ το παρόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάντερ Κάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν γνωρίζω το ιστορικό. Καταλαβαίνω βέβαια αυτά που μας <clears throat> περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι κάνει τώρα. Αλλά πότε τελικά θα εισαχθεί το σύστημα και πότε θα γίνει υποχρεωτικό. Θα είναι οδηγία ή όχι. Το βασικό είναι πότε θα θεσπιστεί το σύστημα και Ποιο θα είναι το κόστος όχημα. Έχετε κάποια ιδέα. Θα είναι δαπανηρή η εισαγωγή αυτού του συστήματος. Δεύτερον, κάνουμε κάποια πειράματα τύπου πλατούνινγκ. Δηλαδή, βάζουμε το ένα φορτηγό, την μια πίσω από την άλλη, δημιουργώντας ε, ένα τέτοιο αεροδυναμικό σειρμό. Ε, αυτό το αεροδυναμικό τούνελ που θα δημιουργήσει το πλατούνι και αυτή η διάταξη στη σειρά των φορτηγών, τι αποτέλεσμα θα έχει στην κυκλοφορία. Και επίσης, ε, τι γίνεται με τις ε, βαριές δαλίκες μεγάλου μήκους. Γιατί μιλήσατε για τις συνδυασμένες μεταφορές. Ισχύει αυτό και για τα, τις μεγάλες δαλίκες με τα ρημολκούμενα. Ναι. <coughs> Μάιλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωί. Και εγώ θέλω, ο γιος Ερτούγμα, ε. θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τις εξηγήσει τη. Όσοι ήταν παρόντε και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου ξέρουν την προϊστορία του θέματος αυτού και τα πολιτικά προβλήματα. Η πλειοψηφία τότε ήθελε όσο δυνατόν να μεταφέρει την μεταφορά φορτίων από το δρόμο στα, στο σιδηρόδρομο. Και επομένως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μπορούν αυτά τα φορτηγά οχήματα να φορτώνονται στο σιδηρόδρομο χωρίς προβλήματα. <coughs> και αυτό είναι το, είναι και το πρόβλημα γιατί αυτή η μικρή φράση που ανέφερε η Κομισιόν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα περιορισμό της δυνατότητα μεταφόρτωσης των φορτηγών στα σιδηροδρομικά βαγόνια. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα πράγματα όπως έχει αποφασιστεί στον Τρίλογο και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο και εκεί ακριβώς έγινε η διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου <clears throat> και Κοινοβουλίου. Το αν είναι αφαιρέσιμα ή όχι αυτά τα, αυτοί οι εξοπλισμοί δεν είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να υπάρχει δυνατότητα όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα στην Ευρώπη να μπορούν να φορτωθούν σε βαγόνια. Ευχαριστώ. Η Γκεζίνε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ασχοληθήκα άμεσα με το θέμα αυτό και μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν αφορά τα μακρύτερα φορτηγά, αφορά τα κανονικά φορτηγά γιατί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φορτώνονται ασφαλώ σε βαγόνια και συγχρόνως να επωφελούνται των καλύτερων αεροδυναμικών συνθήκων. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φορτηγά αυτά στην, στις συνδυασμένες ε, μεταφορές. Σε φυσιολογικές συνθήκες αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μοντέλα που έχουμε δει με πρόσθετα πτερίγια δεν μπορούν να φορτωθούν σε βαγόνια. Αλλά είδαμε στη Γαλλία και στις Ηνωμένε Πολιτείες ότι ορισμένα αυτά μπορούν πράγματι να μεταφερθούν από βαγόνια παρά το γεγονός ότι έχουν αυτόν τον εξοπλισμό. και υπάρχουν ήδη στη Γερμανία, στη, στο Facebook, ε, εξελίξεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε τέτοια φορτηγά τα οποία μπορούν να, ε, να εγκατασταθούν σε βαγόνια. Νομίζω ότι αν έχουμε τη δυνατότητα όμως την τεχνική να μεταφέρουμε περισσότερα φορτηγά από το δρόμο στο σιδηρόδρομο, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε μια τέτοια κίνηση, εγώ νομίζω το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα της συνδυασμένης μεταφοράς και τα άλλα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε με πραγματιστικό τρόπο. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω, είμαι κάπως αδίμονη πόσο καιρό θα κρατήσει ώστε να γίνει αυτή η ρύθμιση, αυτό είναι το θέμα, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί αυτή η, η πρόταση. Κρίμα που δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα το πιο γρήγορα. Αναρωτιέμαι γιατί καθυστερεί όλα, όλη αυτή η διαδικασία. Η ελπίδα μου είναι ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Πότε θα έχουμε τη μελέτη όμως για τα φορτηγά, πότε θα μπουν αυτά τα νέα φορτηγά στον δρόμο και πότε θα μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε σε συνδυασμένες μεταφορές. Ευχαριστώ. Κοίτα Λούγκεν. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ δεν βλέπω που έγινε το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να προσθέσουμε τέτοιου είδους οπίσθια πτερίγια. Έχουμε φορτηγά ήδη με δύο εμπορευματοκιβώτια ρημουρκούμενα και που φέρουν τέτοιο σύστημα οπίστιων αεροδυναμικών συστημάτων. Και μάλιστα είναι πιο εύκολο να προσθέσουμε οπίστη πτερίγια παρά στο μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ίσως ε, αν έχουμε φορτηγά με των 11 τόνων θα έχουμε πρόβλημα ε, γιατί χρειαζόμαστε μοχλούς ε, που να μπορούν να σηκώνουν τόσο βαριά φορτηγά για να προσθέσουν αυτά τα οπίστια πτερίγια. Επίσης, να, προσέξουμε, να προσέξουμε πως δημιουργηθεί υπερβολική πίεση στον κινητήρα. Επίσης, ε, στην εκφόρτωση ίσως δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και στη φόρτωση. Πέραν τούτου δεν υπάρχει πρόβλημα και ο κανόνας των 20 εκατοστών δεν δημιουργεί για μας πρόβλημα. Τεχνικά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν δυσκολίες. Ήδη έχουμε τέτοιε λύσει. λύσεις. Ο κύριος Ζέμκε. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο συνάδελφος. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχαμε συζητήσει αυτές τις αλλαγές και θυμάμαι ένα βασικό στοιχείο ήταν να αποφύγουμε την ε, υπερβολική φόρτωση του οδικού δικτύου και να μεταφέρουμε ένα τμήμα των εμπορευματικών μεταφορών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και από τη μια οι παραγωγοί πιέζουν για να αυξήσουν την παραγωγή των φορτηγών όσο γίνεται και μάλιστα μερικοί το κάνουν, αλλά νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ρέει απρόσκοπτα ε, η μεταφορά και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει αυτά τα πρότυπα και προδιαγραφές να διευκολύνουν την ροή στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Επίσης, ε, δύο νομικά θέματα, γιατί υπάρχει μια σάφια κατά τη γνώμη μου. Αυτές οι νομικές πράξεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα νέα, τα καινούργια φορτηγά και αν ναι, πότε θα προβλέψουμε την προσαρμογή των παλιών φορτηγών, των εκατοντάδων χιλιάδων φορτηγών που ήδη κυκλοφορούν. Είναι θέμα χρονικό, γιατί έχουμε φυσικά την κατασκευή νέων φορτηγών και την παραγωγή νέων φορτηγών, αλλά τι θα γίνει με τα παλιά. Θα προβλέψουμε ένα χρονικό διάστημα για την προσαρμογή τους. Τέλος, από αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κατάλαβα ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες ε, οι νομικές πράξεις. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δοκιμές ώστε η έγκριση τύπου και οι όροι χρήσης ε, να συμπεριληφθούν στην ίδια νομική πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος. Έβαλα τον εαυτό μου ως τελευταίο στο κατάλογο Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να περάσει τη δυνατότητα κυκλοφορίας των μακριτέρων φορτηγών με μια τεχνική προσαρμογή ή οτιδήποτε, μια ερμηνεία. Γι' αυτό νομίζω ότι όλα αυτά ήταν ένα τέχνασμα ώστε μέσω ναι. της αεροδυναμικής αυτής ε, δυνατότητας προσαρμογής να εγκριθούν τα μεγαλύτερα φορτηγά στους δρόμους. Μήπως λοιπόν αυτό είναι απλώς ένας τρόπος για να παρακαθούν τα, η απαγορεύση των μακριτέρων φορτηγών. Αλλά ο Τρίλογος κατέδειξε ότι δεν ήταν αυτό το θέμα και τελικά <clears throat> το θέμα ήταν να μπορεί να υπάρξει αυτή η οριακή επιμήκυνση κατά 20 εκατοστά ώστε να μπορούν να μπαίνουν στα πλοία και στο σιδηρόδρομο τα φορτηγά αυτοκίνητα. Αυτό ήταν αυτό λοιπόν το οποίο θέλαμε να εξασφαλίσουμε. Αυτό το οποίο δεν κατάλαβα και το βλέπω πρώτη φορά εδώ σε 11 χρόνια στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, η Κομισιόν <coughs> μέσα στη διάρκεια ενός τριλόγου να αλλάζει κατά 180 μοίρες πορεία. Έχουμε κάνει πολλούς τριλόγους, έχουμε καταλήξει σε πολλές συμβιβαστικές λύσεις που μπορεί να μην μας αρέσουν ως άτομα. Αλλά όταν τελείωνε η διαδικασία δεχόμασταν το αποτέλεσμα. Από τη δική σας πλευρά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι υπήρξαν πολλά σοβαρά ασφαλότητα από τη δική σας πλευρά. Αν ήταν εδώ ο κύριος Λάιφτριτ, θα σας τα έλεγε λιγάκι πιο χήμα νομίζω αλλά τώρα είναι βέβαια υπουργό <coughs> μεταφορών σε ένα μοσποδιακό κρατήδιο τη Αυστρία. Εμεί ε, ακολουθούμε τη θέση του κ. Λάιχτφριντ, ο οποίο ήταν εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου στον Τρίλογο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη για την Επιτροπή σχετικά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Καταρχήν αυτά, αυτός ο εξοπλισμός που δεν είναι, υποχρεωτικός. Αυτό που λέει οδηγία είναι ότι προβλέπεται εξαίρεση για την ε, τροποποίηση των μέγιστων ε, διαστάσεων του φορτηγού για να εξοπλιστεί το φορτηγό όσων το επιθυμούν. Είτε πρόκειται για νέα είτε για παλιά φορτηγά. Ισχύει εκούσια, θελοντικά το σύστημα. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για προσθήκη αυτών των πτερυγίων. Επίσης, ο δικός μας, η δική μας εκτίμηση αναφέρει 3.000 ευρώ αναφορτηγό. Ε, ρώτησε κάποιος για το κόστος της προσθήκης αυτού του εξοπλισμού. Και θα πρέπει οι μεταφορείς ε, να αποσβέσουν αυτό το κόστος με οικονομία που κάνουν στα καύσιμα, που υπολογίσαμε ότι θα είναι γύρω στο 7% σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση όταν ε, το φορτηγό ε, φτάνει ταχύτητες άνω των 60 χιλιόμετρων, δηλαδή όταν ε, κυκλοφορεί στον αυτοκινητόδρομο ή στους, στις εθνικές οδούς, όχι φυσικά στο εσωτερικό των πόλων. Τώρα για το platooning, για την διάταξη σε σειρά των φορτηγών. Το θέμα είναι βιομηχανικό. Δεν υπάρχει υποχρέωση εξοπλισμού των φορτηγών με το σύστημα αυτό. Οι βιομήχανοι θα πρέπει να πείσουν τους μεταφορείς να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Οπότε είναι προφανές ότι οι όροι χρήσης του φορτηγού, είτε βρίσκεται σε διάταξη είτε όχι, είναι προϋποθέσεις που θα τις εξετάσει ο μεταφορέας για να αποφασίσει αν θα αγοράσει τον εξοπλισμό ή όχι και μπορούμε να μιλήσουμε για το πλατούνινγκ και το αεροδυναμικό τούνελ που θα δημιουργηθεί όταν βάλουμε τα φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο. Πάντως θα πρέπει να γίνουν δοκιμές για τα πτέρυγια αυτά για να δούμε αν βελτιώνουν αυτή τη διάταξη ή αν την παρεμποδίζουν. παρεμποδίζουν τον αεροδυναμικό της χαρακτήρα. Επίσης, θα... δεν ε, βελτιώνει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτό το, αυτό το σύστημα. Αυτό που αναφέρει η οδηγία 719 και ισχύει και για το ε, προστινό μέρος των φορτηγών, οι εξαιρέσεις που αφορούν το μήκος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους μεταφορείς για να αυξηθεί το ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού. Αυτό είναι σαφές. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό ως πρόσχημα για την αύξηση του ωφέλιμου φορτίου. Και ε, ο κανόνας των 20 εκατοστών δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναφέρει στην αγορά ε, πιο μακριά φορτηγά. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Τα rear flaps, αυτά τα οπίστια πτερίγια, μπορούν ε, να εφαρμοστούν στα ΟΜΕΣ, αλλά θα πρέπει να γίνουν πρώτα δοκιμές. Και σίγουρα οι βιομήχανοι θα πρέπει να πείσουν τους μεταφορείς ε, αν θέλουν να προσθεθούν τέτοια πίστια πτερίγια στα φορτηγά. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε το αμπρόστιο ε, από το πίστιο μέρος, γιατί είναι διαφορετικά τα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό η Γενική Διεύθυνση GROW αποφάσισε να διαχωρίσει την ενημέρωση της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στον προστινό από ό,τι στο πίστεο μέρος, γιατί είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα για το εμπρόστιο. Εκεί ανακύπτουν πολλά θέματα. Για παράδειγμα, το βασικό κριτήριο για το εμπρόστιο μέρο είναι ότι χορηγούμε την εξαίρεση μόνο αν η αεροδυναμική απόδοση του φορτηγού βελτιώνεται. Πώ όμω θα καταμετρήσουμε αυτή την αεροδυναμική απόδοση, με τι κριτήρια αναφορά, Όλα αυτά τα συζητήσαμε εκτενώς στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν έχουμε καταλήξει κάπου ακόμη. Όλα αυτά τα θέματα δεν μας προβληματίζουν τόσο για το πίστιο μέρος, για τα οπίστια πτερίγια. Για το, χρονοδιάγραμμα λοιπόν για τα οπίστια πτερίγια είναι... Ε, θα έχουμε την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους όρους χρήσης που θα υποβληθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Τα προϊόντα αυτά σήμερα υπάρχουν στην αγορά ήδη και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες σχεδιάζουν ε, νέα προϊόντα και τα πρώτα φορτηγά που θα εξοπλιστούν με τα συστήματα αυτά θα εμφανιστούν στην αγορά πριν τα τέλη του 2016. Είτε είναι νέα είτε παλιά οχήματα εξοπλισμένα. Για τα παλιά και τα νέα έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα βέβαια. Όσο διαφορά την επικαιροποίηση της έγκρισης τύπου, είπαμε η νομοθετική πράξη θα υποβληθεί μέχρι τα τέλη του 2016, αλλά η οδηγία, όπως ξέρετε, προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για τη θέση σε εφαρμογή των εμπρόσεων αεροδυναμικών συστημάτων. Οπότε, δεχτήκαμε αυτό που μας ζητήσατε να καθυστερήσουμε λίγο περισσότερο για να κάνουμε πιο εκτενείς διαβουλεύσεις. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι η μικρή φράση των 20 εκατοστών καλό θα είναι να διαγραφεί. Κανένα πρόβλημα να διαγραφούν τα 20 εκατοστά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μήκο των φορτηγών. Επουδενή δεν θέλουμε να επαναφέρουμε μακριά φορτηγά στου δρόμου με την πρόταση για τα 20 εκατοστά. Είμαστε υπέρ των συνδυασμένων μεταφορών, ανέκαθεν είμαστε υπέρ των συνδυασμένων μεταφορών και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Και ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις η Γκεζίνη μάλιστα, αν μπορεί να επανέλθει. Αν δεν υπήρξε σφάλμα στην διερμηνία. Νομίζω ότι η Κομισιόν ανέφερε ότι ανέφερε στα οικολογικά ε, φορτηγά, τα οποία είναι μια φορτισμένη εν και πολιτική κρίση σε σχέση με τα οχήματα. Αυτό δεν πρέπει να το πολιτικοποιεί πολύ. Και εγώ, εγώ χάρηκα που το λες αυτό γιατί και εγώ θεώρησα ότι είναι κάποιο πρόβλημα γιατί άκουσα να λέει η Κομισιόν τα monster trucks τα οποία δεν είναι ακριβώς τα οικολογικά ε, φορτηγά. Εντάξει. Εντάξει, ναι, ναι, όχι, δεν φταίει η Κομισιόν, αυτό ήταν απλώς λανθασμένη μετάφραση, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ σύντομα, αν θέλετε να πείτε κάτι, ναι. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Γκόλνης. Έχω δύο διαδικαστικά και δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο διαδικαστικό είναι ότι είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη αυτού του κοινοβουλίου. Παλαιότερα στις επιτροπές σερβιριζόταν καφές ή τσάι. Και πιστεύω πως είναι λυπηρό που δεν έχουμε, γιατί εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να δουλέψουμε, αλλά τα μπαρ και τα καφενεία του κτηρίου είναι κλειστά. Δεύτερη παρατήρηση, ε, στην πολιτική μου ζωή ήμουν νομικός και ήμουν 10 χρόνια μέλος της νομικής επιτροπής. Βρίσκω ε, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφραστούμε για διατάξεις που θα τροποποιήσουν οδηγίες, ενώ δεν έχουμε σχεδόν ποτέ το κείμενο της οδηγίας που υποτίθεται ότι πρέπει να τροποποιήσουμε. Δηλαδή το θέμα της κωδικοποίησης ε, του ευρωπαϊκού δικαίου είναι λίγο κοινό τόπο. Έρχεται και επανέρχεται. Εγώ πάντω δεν μπορώ, δεν μπορώ να πάρω θέση για ένα κείμενο ε, και να τροποποιήσω ένα άλλο εφόσον δεν έχω το προηγούμενο κείμενο. Και τελευταία μου παρατήρηση εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία γιατί πριν από κάποια χρόνια είχα συναντήσει έναν Γάλλο γερουσιαστή που ήταν επικεφαλής μιας πολύ σημαντική επιχείρησης με μεταφορών, οδικών μεταφορών, αλλά γενική φύσης παρατήρηση που ήθελε οι διατάξει για το μάκρο των φορτηγών να ισχύει για το εφόλυμο φορτίο και όχι για το σύνολο του φορτηγού. Γιατί αν μετρήσει κανείς ένα φορτηγό σε όλο του το, τις διαστάσεις, το αποτέλεσμα είναι ότι ο κατασκευαστής μειώνει στο μήνυμο το μέγεθο τη καμπίνας του οδηγού για να αυξήσει όσο γίνεται το φέλιμο φορτίο και αυτό προκαλεί πολλά ε, και ακόμα και θανάσιμα ατυχήματα. Γιατί σε σχέση με το τι κάνει, ε, κάνουν στη ΣΥΠΑ, η καμπίνα ε, δεν προστατεύεται αρκετά στην Ευρώπη και παίρνει όλο το σοκ σε περίπτωση σύγκρουσης οδηγός. Ευχαριστώ πολύ. Να πω το εξής ο καφές και το τσάι έχει σταματήσει να σερβίρεται γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι καφετέρες οι οποίες ε, παραμένουν ανοιχτές, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Για το έγγραφο τώρα που είπατε, το έγγραφο αυτό έχει αποσταλεί, αλλά ίσως για κάποιο λόγο δεν το έχετε λάβει εσείς. Ίσως ε, μπορείτε να το ζητήσετε από την Κομισιόν για να το διαβάσετε. Και τώρα. Σας ευχαριστώ την Κομισιόν για τη συζήτηση και την παρουσίαση. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η, ο έλεγχος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Κομισιόν για τα μέτρα που αφορούν την αεροπορική, ε, τον αεροπορικό κλάδο, εξέταση και περιοδικός έλεγχος πιλότων αποφυγή ενέργειας σύγκρουσης πιστοποιητικό παρόχων υπηρεσιών δεδομένων. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει αυτές τις ε, τρεις προτάσεις για τον έλεγχο και το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εγείρει αντιρρήσεις για τα θέματα αυτά σε σχέση με τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πρόταση για τα συστήματα αποφυγής συγκρούσεων στον αέρα. Ποιος θέλει λοιπόν το λόγο από την Κομισιόν, μπορείτε να αναλάβετε το λόγο για 10 λεπτά αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας και από πλευράς μου. Μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε για διάφορα κείμενα που ήταν στην ατζέντα της τελευταίας ε, συνεδρίας της Επιτροπής ΕΑΖΑ, της Επιτροπής Επιτροπολογίας που επιβλέπει όλους τους εξελιστικούς ε, ε, κανονισμούς που υιοθετούνται υπό τον κανονισμό 216 του 2008 για την ασφάλεια της αεροπλοείας. Τελευταία μας σύσκεψη ήταν τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, και είχαμε διάφορα κείμενα στην ατζέντα μας, όπως σωστά είχατε πει, και αυτά τα κείμενα δεν είχαν ακόμα υποβληθεί όλα για έλεγχο στο Συμβούλιο και την, το, το Κοινοβούλιο, διότι δεν ολοκληρώθηκαν οι συζητήσει σε όλα αυτά τα κείμενα. Όπω θα δείτε από τη σύνοψη των πρακτικών ε, της ε, σύσκεψης αυτής που εντωμεταξύ έχουν ανέβει στο Μητρό, στο έχουν καταχωρηθεί. Το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι η τροποποίηση του κανονισμού 1178 του 2011 που είναι ο κανονισμός που αφορά τον, την, την άδεια πιλότου και το πλήρωμα. Εδώ λοιπόν συνήθως περιλαμβάνονται γίνονται κάποιε αλλαγέ οι οποίε δεν σχετίζονται άμεσα η μία με την άλλη. Γιατί τώρα που έχουμε συστήσει όλου του βασικού κανονισμού για τον έλεγχο των πιλότων, για τα αεροδρόμια, για τα πληρώματα, προσπαθούμε να τι τροποποιήσουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ε, ώστε να είναι ενήμερε, αλλά να αποφεύγουμε να ενημερωνουμε τρει τρει-τέσσερι φορέ το χρόνο. Γι' αυτό και οι αλλαγέ που γίνονται πολλέ φορέ δεν έχουν σχέση μεταξύ του. Τώρα, εδώ στην 1178 ε, οι βασικέ αλλαγέ αλλαγές αφορούν την προσαρμογή της κατάρτισης των πιλότων μέσω του εξυγχρονισμού της αεροπλοείας, ε, αεροπλοήγησης, ώστε να εισαχθούν ε, στοιχεία που βασίζονται στην ε, πλοήγηση με βάση την απόδοση. Αυτό είναι απαραίτητο για τους πιλότους που έχουν μια ταξινόμηση για την, ε, για τις επιδόσεις και για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το BBN, όπως λέγεται στην ορολογία της ε, αεροπορίας. Επίσης, ε, για τους πιλότους που ήδη έχουν αξιολογηθεί για τη χρήση των μέσων, θα μπορούν να αξιολογηθούν για τη χρήση του προνομίου BBN, όπως αποκαλείται γίναν διάφορα αιτήματα για αποσαφήνιση του κειμένου στην τελευταία συνεδρίαση, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει στη διάρκεια της συνεδρίασης και γι' αυτό μετά τη συνεδρίαση υποβάλαμε το κείμενο σε ψηφοφορία δια της γραπτής διαδικασίας και μόλις αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Με θετική γνωμοδότηση, ώστε το κείμενο θα έρθει στις αρχές του επόμενου χρόνου εδώ για έλεγχο. Το δεύτερο κείμενο που είχαμε να εξετάσουμε ήταν ε, μια τροποποίηση στον κανονισμό OPS 965 του 2011. Επίσης και πάλι ε, με κάποιες αλλαγές στο PBN, κάποιες αλλαγές επίσης για τους παρόχους υπηρεσιών δεδομένων, ε, ε, επίσης το πώς μαθαίνουμε από τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και κάποιες διορθώσεις ε, διατύπωσης. Τέσσερις διαφορετικές ονομοδοτήσει ε, της ΕΑΖΑ οδηγούν σε αυτές τις τροποποιήσεις του κανονισμού 965. Αυτό το κείμενο στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής δεν ήταν ε, πίμαχο εκτός από ένα σημείο όπου επιφέραμε μια αλλαγή στην προσέγγιση της εισαγωγής νέων κανόνων. Στο παρελθόν συχνά για αυτούς τους κανονισμούς είχαμε περιόδους opt-out όπου κάποιο κράτος μέλος θα μπορούσε μονομένα να αποφασίσει ότι θα ε, δεν θα συμμετέχει για μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως δύο, ε, διάρκειας δύο ετών. Στο παρελθόν όμως είχαμε προβλήματα, γιατί τότε η κατάσταση δεν ήταν ίδια στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπήρχαν ζητήματα σαφήνειας για το ποια είναι η κατάσταση, ζητήματα αμοιβαίας αναγνώριση και αποφασίσαμε να αλλάξουμε αυτή την προσέγγιση ώστε τα opt-out να ξεκινούν σε κοινέ ημερομηνίε εφαρμογή για όλα τα κράτη-μέλη. Βασικά δηλαδή ισχύει το opt-out για όλους τώρα. Τώρα, επειδή ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό, διάφορα κρατημέλη είπαν πως αυτό τους δημιούργησε προβλήματα. Η μετάβαση από τους παλιούς κανόνες στους νέους, γιατί στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν το opt-out για να εκδώσουν νέες άδειες επί τη βάση των νέων κανόνων, αλλά ακόμα και αν είναι οι κανόνες δεν ήταν απόλυτα εφαρμοστέοι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρακτικά ζητήματα Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το διορθώσουμε στο κείμενο και θα επανέλθουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας που νομίζω είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο με λύση ε, για αυτό το νομικό πρόβλημα της μετάβασης. Και βέβαια σε περίπτωση θετικής νομοδότησης θα έρθουμε εδώ στο Κοινοβούλιο μάλλον τον Μάρτιο. Το τελευταίο κείμενο τώρα που ήθελα να σας αναφέρω είναι η τροπολογία στον κανονισμό 1332 του 2011 ειδικό κανονισμός για την αποφυγή εναέρειας σύγκρουσης. Και εκεί κάναμε αλλαγές επί τη βάση της νομοδότησης υπαριθμών 4 του 2014 της ΕΑΖΑ το κείμενο αυτό δεν ε, ήταν επίμαχο, ήταν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν εδώ αρκετές, ε, αρκετά σημεία για το κανόνες του ενιαίου ουρανού που το διαχειρίζεται μια άλλη επιτροπή. Το κείμενο αυτό λοιπόν συμφωνήθηκε και πιστεύω πως εστάλει στο Κοινοβούλιο για έλεγχο μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ποιος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Μπάχ, ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε. Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για μένα. Και έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε χάσει κάποιο χρόνο. Αλλά δεν φταίμε εμείς γιατί δεν είχαμε όλα τα κείμενα στα χέρια μας και θα πρέπει να αναζητήσουμε το χαμένο χρόνο μέσα από τα έγγραφα. Είναι καλό λοιπόν τον Φεβρουάριο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν προβλήματα με αυτή την αυτοεξαίρεση, το opt-out των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα τι περιέχουν τα κείμενα αυτά και να ασχοληθούμε και με την ε, θέση των εθνικών κρατών, ώστε να υπάρξει μια κάποια συμφιλίωση μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω καταλάβει τη στιγμή πού βρίσκονται οι δυσκολίες φυσικά ή αν αυτά είναι απλώς προσχήματα για να καθυστερήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ την Κομισιόν. Ένα ερώτημα για την εκπαίδευση των πιλότων προβλέπετε ή εξετάζετε; Να μπορούνε να πετούντα αεροπλάνα μένα φιλότομονάχα. Ξέρω ότι σπεύσονται σε φορές πετάνε αυτόματα τα αεροπλάνα. ή εξεταζετε να μπορούν να πετούν τα αεροπλάνα με ένα πιλότο μονάχα. Ξέρω τις περισσότερες φορές πετάνε αυτόματα τα αεροπλάνα. Η, η τεχνολογία βέβαια γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και αναρωτιέμαι αν οι πιλότοι πραγματικά είναι σε θέση να παρακολουθήσουν όλη αυτή την πολυπλοκότητα της ε, τεχνολογίας. Είναι σε θέση λοιπόν οι πιλότοι να χρησιμοποιούν πραγματικά και να διαχειρίζονται όλα, όλη αυτή την τεχνολογία η οποία βρίσκεται εγκαταστημένη στα cockpit. <coughs> Νομίζω λοιπόν ότι έχει φτάσει να είναι σαν διαστημική πτήση το να πετάει κανείς σε ένα αεροπλάνο και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κ. Ευχαριστώ. Το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που σας είπα και προηγουμένως και με παρεξηγήσατε νομίζω. Σας είπα ότι συζητούμε αδιάκοπα κείμενα που τροποποιούν οδηγίες ή κανονισμούς, στους οποίους δεν έχουμε λάβει, δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Και άρα δεν είμαστε κατατοπισμένοι. Μας είπατε ότι μοιράστηκαν τα έγγραφα. Μα Διάβασα και μάλιστα ενδελεχώς τα έγγραφα που μοιράσατε, αλλά γιατί πράγμα μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ένα νέο κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό 1332 του 2011. Για παράδειγμα διαγράφει το άρθρο 4. Ο συνάδελφος εδώ που γνωρίζει τι προβλέπει το άρθρο 4 του κανονισμού 1332 που προτείνεται να καταργηθεί. Νομίζω ότι κανείς δεν το γνωρίζει θα πρέπει ο καθένας να ψάξει μόνος του. Εγώ, παρόλο που είμαι νομικός, αδυνατό να συζητήσω για ένα κείμενο που τροποποιεί προηγούμενο κείμενο το οποίο δεν έχω στη διάθεσή μου. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Αν όμως όλα αυτά μα τα είχατε εξηγήσει, τα μοιράσει εκ των προτέρων, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Να είχαμε αμύτη άλλο μπροστά μα το κείμενο του άρθρου 4 που θέλετε να τροποποιήσετε, να καταργήσετε. Εγώ δεν είμαι νομομαθής, αλλά συμφωνώ μαζί σας και εγώ δεν μπορώ να συζητώ για κείμενα τα οποία δεν ξέρω τι λένε. Αλλά στο έγγραφο της ε, κομιτολογής σε όλες τις γλώσσες υπάρχει το κείμενο αυτό και μπορούν οι βουλευτέ να το διαβάσουν. Άμα δεν θέλει κανείς να το διαβάσει, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε ότι δεν έχετε διαβάσει το κείμενο γιατί δεν υπήρχε. Μπορείτε να το βρείτε εκεί και στην γλώσσα σα. Και εγώ έχω ένα ερώτημα προ την Κομισιόν, ο κ. Σέτου. Γιατί ακριβώ και αυτό το θέμα συζητούμε πριν από δύο εβδομάδε στο Σπίγκερ, στο γερμανικό τύπο, αναφέρθηκε ότι σε σχέση με το ατύχημα της ε, German Wings το Μάρτιο, οι γερμανικές ενώσεις πιλότων θέλουν να υπάρχουν ευνηδιαστικοί έλεγχοι στους πιλότους για χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν γνωρίζει αυτά τα σχέδια στη Γερμανία και αν έχει μια θέση για τα θέματα αυτά και εγώ θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα μετά το ατύχημα της German Wings. Τι ακριβώς έχει γίνει για να αντιμετωπίζονται τα ψυχολογικά προβλήματα των πιλότων. Τι γίνεται για να αντιμετωπιστεί η κόπωση των πιλότων. Πού τίθενται τα όρια στην αντοχή των ανθρώπων αυτών και επίσης το θέμα της ποιότητας της, ε, του αέρα της, ε, ε, του πιλωτήριου. Γιατί υπάρχει περίπτωση πιλότων που έχουν αποκοιμηθεί γιατί ήταν πραγματικά τοξικό το περιβάλλον της, ε, του πιλωτηρίου. Πώς μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό της, ε, του, της ατμόσφαιρας στο πιλωτήριο που δεν αφορά φυσικά μόνο τους πιλότους αλλά και τους επιβάτες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σχόλιο για τις ημερομηνίες και πότε διατίθεται τα κείμενα. Καθυστέρησαν τα κείμενα δεν είναι ότι εμεί καθυστερήσαμε. Εσεί πέψατε να θέσετε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εσεί παρέσασταν ναι. γρήγοροι. Και σε δύο από τα τρία κειμένα δεν έχει καν ψηφίσει η Επιτροπή. Μόνο πριν από λίγε μέρε ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για ένα από τα τρία κείμενα. Και μόνο μετά τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Επιτροπολογία μπορούμε να στείλουμε το κείμενο. Τα υπόλοιπα δύο κείμενα θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιτροπολογίας. Και τότε θα γίνει η ψηφοφορία το νωρίτερο στην επόμενη τη συνεδρίαση. Τώρα, για την εκπαίδευση των πιλότων και πώς ε, πρέπει να συνδυάζουμε την εκπαίδευσή τους ε, με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Άλλο τα μεγάλα αεροσκάφη, ε, και οι πιλότοι εκπαιδεύονται και συγκεκριμένα είδη αεροσκαφών που γίνονται όλο και πιο εξεζητημένα και άρα η εκπαίδευσή τους προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες. Και αυτό αποτελεί τμήμα της πιστοποίησης των αεροσκαφών. Δίνονται στην πιστοποίηση ενδείξεις για την απαιτούμενη εκπαίδευση του πιλότου, ώστε να συνάδει με το, τον τύπο και τη λειτουργία του αεροσκάφους. Εδώ όμως μιλούμε κυρίως για μικρότερα αεροσκάφη και πιλότους ε, ιδιώτες, ιδιωτικά αεροσκάφη και έτσι εκεί χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλοήγηση βάσει βαση επιδοσεων το PMB, όχι παντού ταυτόχρονα βέβαια στον αέριο χώρο, εξαρτάται και από το αεροδρόμιο. Εκεί που ισχύει όμως, οι πιλότοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε τέτοιο περιβάλλον. Οπότε και η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένη και να παρακολουθεί την πρόοδο στις τεχνικές πλοήγησης. Για το τελευταίο σημείο, τους ελέγχους ε, για χρήση ναρκωτικών και ενοπνεύματος δεν το συζητήσαμε στην Επιτροπή της ΕΑΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας. Η ΕΑΣΑ μάλιστα θέσπισε και σχέδιο δράσης μετά την ε, συντριβή του αεροσκάφου της German Wings και μάλιστα το σχέδιο δράσης βρήθη καλών προτάσεων και ιδεών, πρέπει όμως να εξεταστούν ενδελεχώς ε, και από εμπειρογνώμονες για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν στην πορεία και αν θα οδηγήσουν σε νομοθετικές αλλαγές ή απλώς ε, σε συστάσεις. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια του 2016. Οπότε θα επανέλθουμε μετά την κατάθεση των προτάσεων. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα στο πιλωτήριο ή στην καμπίνα του αεροσκάφους, δεν είναι κάτι καινούριο βρίσκεται υπό έλεγχο και μάλιστα είχαμε τέτοια κρούσματα ε, σε, στο συγκεκριμένο, και το αναφέραμε στο συγκεκριμένο κανονισμό και μάλιστα τώρα υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης για να δημιουργήσουμε καλύτερη εικόνα τέτοιου είδους ε, περιπτώσεων και μάλιστα η ΆΣΑ συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα για την εξέταση αυτού του θέματος, γιατί ακόμη ε, τα επιστημονικά πορίσματα δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Και το θέμα της κόπωσης των πιλότων. Οι νέοι κανόνες για τον περιορισμό των ορών πτήσης, ε, που δεν είναι και πολύ ε, παλιές, θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Οπότε όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις για τον περιορισμό των ορών πτήσης. Αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός, που στόχο έχει να ελαφρύνει αυτό το θέμα της κόπωσης. Ωραία, λοιπόν. Οι προθεσμίες για τη διατύπωση αντίρρησεων 28 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την Επιτροπή μας και 1η Μαρτίου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Παίρναμε τώρα στην ακρόασή μας για την ε, αεροπλοεία και θα ήθελα να παρακαλέσω τους ομιλητές να λάβουν τις θέσεις τους.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 So, Έχουμε έξι ομιλητέ. Θα του παρουσιάσω όταν λαμβάνουν το, το λόγο. Θα ακολουθήσει λοιπόν συζήτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σα Για να ασχοληθούμε με το θέμα του ανταγωνισμού στην διεθνή αεροπλοεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κλάους Γκάιλ από την DG Move. Συγγνώμη, συγγνώμη. τον κύριο Λαμπρόσο από το Διεθνές Φόρουμ του Μεταφορών του ΟΣΑ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμπρόσο. Mr. Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable parliamentarians, ladies and gentlemen. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτέ, είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σα μιλήσω λίγο από τη δική μα προοπτική για τον ανταγωνισμό στη διεθνή αεροπλοεία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομάζομαι Αλέν Λαμπρόζο, είμαι οικονομολόγο στο Διεθνέ Φόρουμ για τι Μεταφορέ του ΟΑΣΑ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά την Γραμματεία και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ και να υπογραμμίσω την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που έκανε η Κομισιόν πριν κάνει την πρότασή της για την αεροπλοεία. Ε, πραγματικά ήταν πλήρης ε, ε, πληροφοριών, μας χαροποίησε όταν τη διαβάσαμε και ελπίζω πως θα σας διαφωτίσουμε για το πώς βλέπουμε την κατάσταση. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Σύντομα λοιπόν για το τι είναι αυτό το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών. Είμαστε μια διακυβερνητική οργάνωση με 57 χώρες μέλη, 27 από την Ένωση. Δεν μιλάμε εξ ονόματος των χωρών μελών μας, είμαστε ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός Ανάμεσα σε αυτά που κάνουμε είναι ότι έχουμε την λειτουργία της ε, δεξαμενής σκέψης, think tank, ε, ας πούμε ενημερώνουμε και δίνουμε τις γνώμες μας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης λειτουργούμε το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Σύστημα Ποσοστώσεων για την ανείχνευση και την παρακολούθηση, αλλά και φιλοξενούμε το, τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής Υπουργών μεταφορών στην Γερμανία που συμμετέχουν και οι Υπουργοί της Ένωσης. Ήδη γνωρίζετε τα γενικά στοιχεία για την, ε, την αεροπλοεία. Είναι τεράστια βιομηχανία, 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, αλλά φυσικά ο αντίκτυπος, ο πραγματικός δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι και η διασύνδεση, η κινητικότητα, είναι αυτός ο ιστός των διεθνών οικονομικών μας οργανισμών. Ωστόσο, βλέπει κανεί την αεροπλαία εντό τη Ένωση, διαπιστώνει ότι το κέντρο ε, βαρύτητας μετακινείται προς Ανατολάς, προς τα ανατολικά σύνορα τη Ένωση και πέρα από την Ένωση προς την Ασία περισσότερο. Οπότε αυτό που συμβαίνει και αυτό που βλέπουμε εδώ στα δεξιά, από το 2008 μέχρι το 2014 είδαμε ανάπτυξη στην ε, μεταφορά επιβατών στην Ευρώπη αλλά ξεκινάμε από πολύ μικρότερη ε, βάση. Αναπτύσσεται η κίνηση στην Ευρώπη, αλλά όχι όπως αλλού εντός της Ευρώπης και γύρω από τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, έχουμε λοιπόν προβλέψεις για την ε, κίνηση, μετακίνηση επιβατών. Είμαστε στο 10% της παγκόσμιας αγοράς και αυτό που αναμένουμε μέχρι το 2030 είναι μεγάλη αύξηση στην Ευρώπη. Θα διπλασιαστεί μάλιστα η κίνηση και αυτό δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει με την ανάπτυξη που θα δούμε στον υπόλοιπο κόσμο που είναι γύρω στο 140% ή ακόμα και τριπλασιασμό στην Ασία και την Αφρική. Άρα λοιπόν η ε, αεροπλοεία αυξάνεται, αυξάνεται στην Ευρώπη, ε, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε το, το μερίδιο της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώνεται όσο πάει. Και αυτό είναι, οφείλεται σε διάφορους μακροοικονομικούς, κοινωνιολογικούς και δημογραφικούς λόγους και δεν συνδέεται συγκεκριμένα με την πολιτική μεταφορών. Η ε, αεροπλοεία θα διπλασιαστεί ωστόσο στην Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τα θέματα ας πούμε, της συμφόρησης των αεροδρομίων, του, ε, ε, τη συμφόρηση του ενάριου χώρου και πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτά, τις δομές που έχουμε ή αλλιώς να εξασφαλίσουμε ε, τις δομές για τη μελλοντική ζήτηση. Θα έρθει. Τώρα, όταν κανείς εξετάσει το διεθνή ανταγωνισμό στην αεροπλοεία, ένα από τα πρώτα πράγματα που διαπιστώνει στο πρόγραμμα το ερευνητικό είναι το επίπεδο, ε, το ισότιμο πεδίο για όλους. Όλοι είναι υπέρ, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς υπέρ πρόκειται. Έχουμε 45, 40 ε, μάλλον ειδικού σε μια αίθουσα ε, και δεν συμφωνούν μεταξύ τους για το τι είναι το ισότιμο πεδίο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα σε ε, κάποιες επικράτειες, ενώ άλλα σε άλλες. Όταν δούμε όμως τη σύμβαση του Σικάγου, μιλάει για ισότητα ευκαιριών, αλλά όχι για ισότητα ε, ε, αποτελεσμάτων ή επιδόσεων. Άρα σημαίνει αυτό πως κάποιοι μεταφορείς έχουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με το ισότιμο πεδίο εξ αρχής, αλλά και τη διαχείριση αυτού. Αυτό εδώ το γράφημα που βλέπετε το έχουμε βουτήξει από τη Λουφτχάνσα ε, χωρίς πολλά πολλά, αλλά είναι ένα εξαιρετικό γράφημα που δείχνει ότι ε, όσο περισσότερο απ' έξω είσαι, τόσο πιο εύκολο είναι το περιβάλλον, τους, το περιβάλλον σου, λειτουργία σου και όσο πιο μέσα είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι. Η Λουφτχάνσα είναι ο κίτρινος κύκλος και ο μπλε κύκλος είναι η, τα Εμμυράτα. Ναι. Ε, και αυτοί λειτουργούν πολύ πιο εύκολα, όπως βλέπετε βλέπουμε ότι οι μεταφορείς εντός της Ένωσης και εκτός της Ένωσης λειτουργούν με τελείως διαφορετικούς όρους. Και αυτό και έχει προκύψει αυτή η ιδέα της ισότητας των ίσων όρων που τελικά είναι τελείως θεωρητική όταν δει κανεί ε, πώς λειτουργούν και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι διάφορες ε, αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, κρατικές ενισχύσει. Και αυτό το μελετήσαμε πολύ προσεκτικά. Εντός της Ένωσης είναι πολύ πιεστικές και αυστηρές οι κατευθυντήριε γραμμές για το ποια κρατική ενίσχυση επιτρέπεται και ποια όχι. Και η Κομισιόν έχει προβεί σε διάφορες δράσεις κατά κρατών μελών όταν πίστευε ότι... κάτι πάει στραβά και έχουμε βρει ότι βασικά οι εθνικές κυβερνήσεις θέλουν να έχουν την ελευθερία να παρέχουν κρατικέ ενισχύσει στις εθνικέ του όταν και ε, το κρίνω αυτό απαραίτητο. Το θέμα όμως που υπάρχει εδώ με τις σχετικές ενισχύσεις ε, στη διεθνή αεροπλοεία είναι ότι εκτός της Ένωσης δεν υπάρχει κανένας κανόνας για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο πίνακας που βλέπετε στο δεξί τμήμα της διαφάνειας ε, είναι ένα είναι αυτή η υπόθεση με τον ανοιχτό και δίκαιο ουρανό και το τι λένε τα Εμμυράτα. Δηλαδή, τι θα πει άδικη κρατική ενίσχυση. Ας πούμε, η απαγόρευση στα συνδικάτα, στη, στη ΣΥΠΑ, θεωρείται ε, αυτό κρατική ενίσχυση. Το ότι δεν υπάρχουν τα συνδικάτα λοιπόν θεωρείται είδο επιδότηση. Ενώ στα Εμμυράτα ισχύει κάτι τελείω διαφορετικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο παγκόσμιο καθεστώ ε, για το τι είναι επιδοτήσεις και τι όχι και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν εναντίον ποιου αν δοθούν παράνομα ε, επιδοτήσεις. Ναι, ναι, ολοκληρώνω, ναι. Ε, σε πλαίσιο ΙΚΑΟ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα βασικό ορισμό, ένα κάποιο πλαίσιο του τι επιτρέπεται, πώς καταγράφεται, πώς επαληθεύεται και πώς ε, μπορεί κανείς να προβεί σε μέτρα επιβολής όταν καταβάλλονται επιδοτήσεις που είναι αντίθετες με το βασικό αυτό πλαίσιο. Αλλά λόγω της φύσης της αεροπλοείας αυτό πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο και μόνο η ΙΚΑΟ μπορεί να το κάνει. Δεν ακόμα πολύ πρόοδο πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το επίπεδο. Επόμενη διαφάνεια. Α, συγγνώμη. Α, με συγχωρείτε. Ε, νόμιζα ότι είχα παραπάνω 10 λεπτά. Τρία, τρία δευτερόλεπτα δώστε μου. Όσον αφορά την ε, ιδιοκτησία και τον έλεγχο, ίσως θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε, απελευθέρωση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται από οικονομική πλευρά και όχι από τακτική πλευρά. Επίσης υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο προηγμένη από ό,τι άλλες δικαιοδοσίες στην απελευθέρωση ιδιοκτησίας και ελέγχου. Δύο διαφάνειες παρακάτω, ναι. Ε, βασικά η ιδέα είναι ότι δεν θα έχουμε πραγματικά ίσους όρους στην αεροπλοεία, αλλά είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ανταγωνιστική αγορά που θα έχει πρόσβαση στην διασύνδεση για τους ε, ταξιδιώτες αλλά και για τους ε, μεταφορείς. Θα πρέπει ολόκληρη η αλυσίδα να παραμείνει ανταγωνιστική και ανοιχτή στην αγορά. Τελευταία μου διαφάνεια. Θέλω να σας ευχαριστώ ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω και να σας καλέσω στο συνέδριο τον Μάιο του 2016 στη Γερμανία. Ναι, ναι. Ναι, σας ε, ευχαριστώ. Ναι, όχι 10 λεπτά, 6 λεπτά βέβαια είχατε στη διαθεσή σας. Ακολουθεί ο κύριος Αταρ Χουτσάιν ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος για την Ένωση των Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που με απευθύνετε, Χαίρομαι που μπορώ να είμαι εδώ και να συμμεριστώ μαζί σας μερικές από τις απόψεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών για την κατάσταση ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αεροπλοείας. Αν θα πετάξει τώρα το επόμενο slide δεν το ξέρω. Εντάξει. Να σας δώσω το γενικό πλαίσιο τώρα. Ο συνάδελφός μου προηγουμένως σας έδωσε μερικά βασικά στοιχεία χωρίς να μπούμε σε πολλή λεπτομέρεια. Πιστεύουμε ότι χάρη στην συμπλήρωση της ενίας αγοράς κάτι δεκαετία του 1990 υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, νέες δυνατότητες επιχειρηματικών μοντέλων, ευκαιρίες για τους επιβάτες, ευκαιρίες για τους καταναλωτές, μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Αλλά δυστυχώς τώρα βλέπουμε βλέπουμε ότι μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο ο ανταγωνισμός. Σε άλλες περιοχές του κόσμου βλέπουμε ότι έχουν αναγνωρίσει την αξία της αεροπορίας περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πάρει θεσμικά και οργανωτικά μέτρα. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μια πιο ολιστική αντιμετώπιση της αεροπλοείας, να την αντιμετωπίσει σαν ένα βασικό συστατικό της ε, κοινωνίας μας και γι' αυτό στο στρατηγικό μας σχέδιο ζητήσαμε να εξασφαλίσουμε το ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού. Όπως είπε ο κύριος ο προηγούμενος, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Θα περάσω τώρα σε λεπτομέρειες. Τονίζουμε ότι είναι ουσιαστικό το, ο θεμητός ανταγωνισμός, η ισότητα ανταγωνισμού, ιδίως όταν έχουμε ένα τέτοιο κλάδο και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίο είναι νευραλγικό και πολύ ανταγωνιστικό. Έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να προχωρήσει σε τρία ουσιαστικά βήματα. Να επιβάλλει ρυθμίσει ότι υπάρχει ανάγκη για νομοθεσία για να εφαρμόσει του κανονισμού που ισχύουν, <clears throat> χωρί όμω να υπερφορτώσει την, τον αεροπορικό κλάδο. Με πρόσφατη το άχθος ή πρόσφατο κόστος. Αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε στην Ευρώπη, νομίζω σε μεγάλο βαθμό το εξασφαλίσουμε με αυτορύθμιση. η στρατηγική για, την, για τον αεροπορικό κλάδο που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες τονίζει ότι φυσικά οι αεροπορικές μεταφορές βοηθούν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία, την οικονομική μεγέθυνση, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα και δίνουν ε, εργασία σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα άμεσα ή έμεσα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός συμβολέας στην ε, ευμάρεια και την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η συμβολή του αεροπορικού κλάδου στην οικονομία γενικά αναγνωρίζεται, δεν αναγνωρίζονται οι οικονομικές πραγματικότητες. Ο κλάδος είναι πολύ Ανταγωνιστικό το περιθώριο κέρδους είναι πάρα πολύ μικρό σε αυτόν τον κλάδο. Αυτό το οποίο τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο κατά δική μα άποψη είναι να έχουμε ένα αεροπορικό κλάδο που να εδράζεται στην Ευρώπη και ο οποίο να εξυπηρετεί τα στατηγικά σφαίρα τη Ευρώπη, επενδύσει, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα. Ω παράδειγμα, τονίσουμε ότι οι πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκές εταιρείες ε, δημιουργούν τέσσερις φορές περισσότερη απασχόληση από ό,τι πτήσεις από μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Για να έχουμε λοιπόν ένα δυναμικό τομέα της ευρωπαϊκής αεροπορικού κλάδου. Αυτό δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την ευρωπαϊκή οικονομία και περιμένω από την Κομισιόν να παίξει ένα κύριο ρόλο για τα θέματα αυτά είναι επίσης απαραίτητο να έχουμε και κάποια τάξη που θέσουν, θα θέσουμε στην αγορά. Δεν μπορούμε να δούμε απομεμονωμένα την ευρωπαϊκή αγορά. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε μια πολύπλοκη αλυσίδα προσθέμενης αξίας προμηθευτών και παρόχων. Όταν υπήρξε η φιλελευθερωποίηση, υπήρξε φιλελευθερωποίηση των εταιριών, αλλά όχι του υπόλοιπου τμήματος της αλυσίδας προσθέμενης αξίες. Ξεκολουθούν να υπάρχουν μονοπωλιακοί πάροχοι υπηρεσιών και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας αντιμετώπισης λειτουργούμε σε παγκόσμιες αγορές. <clears throat> Οι Ευρωπαίοι λοιπόν οι μισθές και οι πολιτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν πως τα μέτρα τα οποία θα έχουν πιο άμεσο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σύστημα παραδείγματος χάρη εμπορίας εκπομπών και οι συζητήσεις για το PNR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας δείχνουν παραδείγματα αυτού του προβλήματος. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της εξωτερικής συνιστώσεως των προβλημάτων. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε <coughs> σχέσεις μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξένων χωρών, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του αεροπορικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δώσει ίσες και δίκαιες ε, δυνατότητες ανταγωνισμού. Μας Απογοητεύει λοιπόν το γεγονός ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνει υπόψη την αναθεώρηση του κανονισμού 868 που θα μπορούσε να είναι ένα κομβικό στοιχείο στην επίτευξη των στόχων αυτών. Είναι σημαντικό ο θεμητό ανταγωνισμό, όπω είπε και προηγούμενο ομιλητέ, τα θέματα των κρατικών ε, διασφαλίσεων και των εγγύησεων <clears throat> είναι θέματα που έχουν συζητηθεί και σε επίπεδο ΙΚΑΟ δεν έχουμε φτάσει μέχρι στιγμή σε κοινή συναντήληψη, αλλά υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν για να εφαρμόσει και να προωθήσει τη ρήτρα θεμητού ανταγωνισμού στις διμερείς συμφωνίες, γιατί αυτά είναι τα μόνα εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και έρχομαι στην τελευταία μου διαφάνεια. Πάντα ζητήσαμε να υπάρξει σε αμοιβαία βάση φιλελευθεροποίηση σε σχέση με τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των εταιριών και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και εμεί το ρόλο μα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Τώρα, σε σχέση με την ε, εντολή διαπραγμάτευσης που ζήτησε η Κομισιόν για τρίτες χώρες, τι υποστηρίζουμε, ιδίως με τα κράτη του Περσικού κόλπου, με την ΑΣΕΑΝ, την Τουρκία, το Μεξικό και την Αρμενία. Να κάνω τώρα κάποιες πιο λεπτομεριακές παρατήρησεις. Με τη Βραζιλία διαπραγματευόμαστε από το 2011 και καταλήξαμε σε μια, έπρεπε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το 2011, αλλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Σα δίνω τη Βραζιλία ω ένα παράδειγμα. Όταν η Κομισιόν κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση εξώματο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να είναι ελευκό αυτή η εντολή. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το χρονικό όριζοντα. Υποστηρίζουμε το διάλογο με τα κράτη του Περσικού κόλπου, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών του κόλπου, ακόμα και αν η εντολή αφορά μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες, θεωρούμε ότι ο γενικός διάλογος μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να εξηγήσουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς λειτουργεί η φιλελευθερωποιημένη αγορά και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια αριθμιστική σύγκληση στα θέματα αυτά. Για την Κίνα σιγά σιγά. <clears throat> Πρώτα συμφωνία για την ασφάλεια, μετά η οριζόντια συμφωνία και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για μια πλήρη συνολική συμφωνία. Κάτι το οποίο ξεχωριστώ για την Κίνα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε και ένα πρόβλημα με τις υπερπτήσεις της Σιβηρίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιριών να μην τύχουν ομοιρίας όταν κάνουμε μια συνολική συμφωνία με τους Κινέζους. Αυτό είναι το τελευταίο που ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη που πέρασε το χρόνο μου. Ευχαριστώ και ακολουθεί ο κύριος Τζον Χένλον, γενικός ε, γραμματέας της Ένωσης των Εταιριών Χαμηλού Κόστους. Κύριε Χένλον, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας ε, και σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας. Η ΕΛΦΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αερογραμμών Αυθινών Εισιτηρίων, ε, έχει πολύ ενεργά μέλη, είναι μισή περίπου αεροπορικέ εταιρείε Ευρώπη ε, ενεργοποιούνται και κυρίως στην εσωτερική αγορά. Ορίστε, αυτά είναι τα περισσότερα πιο γνωστά μας μέλη. Φαντάζομαι σας είναι γνωστές όλες αυτές οι αεροπορικέ εταιρείε. Καταρχήν, ποια είναι η γνώμη μας για την αγορά της αεροπορίας. Θεωρούμε ότι η απελευθέρωση είναι σωστός δρόμος ε, δυστυχώς δεν κυριαρχεί παντού αυτή η απελευθέρωση, αυτή η φιλελευθερωποίηση. Έχουμε σημαντική ανάπτυξη εξαιτία της ε, απελευθέρωσης ε, εντός της κοινοτικής αγοράς, κάτι που δεν αντικατοπτρίζεται και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί πολλές χώρες είναι πολύ προστατευτικές των αγορών τους. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απελευθερώσει τις συμφωνίες ασφάλειας της αεροπορίας, έχει ε, περισσότερο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές, φθηνότερα εισιτήρια, περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, χάρη σε αυτή την φιλελευθερωποίηση που έχει επιβάλει. Ποια είναι τα ωφέλη αυτής της απελευθερώσης, αυτής τη φιλελευθερωπής. Καταρχήν ε, βελτιώνεται η συνδεσιμότητα, οι ποιοτικέ ανταποκρίσεις. Αυτό είναι το σλόγγαν ε, της στρατηγικής μας. Πολλά δρομολόγια προσθέθηκαν μετά την απελευθέρωση της αγοράς, κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα τώρα υπάρχουν ζεύγοι πόλων, δρομολόγια που δεν υπήρχαν παλιά, με πολύ συχνές πτήσεις. Η συνδεσιμότητα έχει αυξηθεί κατά 10% που οδηγεί σε 0,5% αύξηση του εθνικού ΕΠ. Είναι αλληλένδετες λοιπόν αυτές ε, οι εξελίξεις ε, ε, αύξηση της συνδεσιμότητας, της απελευθέρωσης και της ανάπτυξης. Αυξάνεται η απασχόληση και πάνω απ' όλα αυξάνεται ο ανταγωνισμός με ε, τους καταναλωτές να βγαίνουν κυρίως κερδισμένοι εξαιτίας της αύξησης των επιλογών και των φθηνότερων εισιτηρίων που μπορούν να βρουν. Ποια είναι τα προσκόμματα στην απελευθέρωση τώρα, στη φιλελευθερωποίηση. Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναπτυχθεί επιτυχώς ε, στην αεροπορία. Έχουμε πολύ καλό ιστορικό, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Τώρα, το θέμα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πρόοδο και στο μέλλον, να συνεχίσουμε την επιτυχία που είχαμε στο παρελθόν. Στο μεταξύ, η αεροπορία ε, έχει γίνει μια παγκόσμια αγορά και οι αγορές εξελίσσονται, αλλάζουν. Οπότε οι παλιές συνταγέ ε, δεν αποφέρουν τους ίδιους καρπούς και την ίδια επιτυχία. Υπάρχει ο φόβος κατά τον αλλαγών πολλές φορές. Κάτι που φαίνεται έντονα σε μερικές χώρες, μερικές χώρες γιατί θεωρούν ότι η απελευθέρωση θα αποδυναμώσει τα συμφέροντά τους και γι' αυτό προσπαθούν να την παρεμποδίσουν ή να δεν επιβραδύνουν. Και μάλιστα λένε κοιτάξτε τι γίνεται με το μερίδιο αγοράς. Αλλά το μερίδιο αγοράς δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύει κανείς. Θα πρέπει να συνεχίζει να το κερδίζει το μερίδιο αγοράς. Δεν είναι ποτέ κεκτημένο και προνόμιο. Επίσης, ε, δεν, είναι, δεν ισχύει η ιδιοκτησία στην εσωτερική αγορά. Δεν ε, είναι ιδιοκτησία κανένα κράτους ε, οι καταναλωτές, οι ταξιδιώτες. Θα πρέπει να είναι ελκυστική η εσωτερική αγορά. Τώρα, ο ανταγωνισμός ενδράσει. δράση. Ακούσαμε πολλά για τον ανταγωνισμό που επιβάλλουν οι χώρες του Περσικού κόλπου. Εμείς Πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι μας βλάπτει δικός τους ανταγωνισμός, αλλά οι δικές τους κυβερνήσεις έχουν μια πολύ πεφωτισμένη προσέγγιση για την αεροπορία. Επενδύουν στις υποδομές, ε, ε, εξεχρονίζουν τα αεροδρόμια, τους διαδρόμους τους και αναπτύσσουν βιομηχανίες που αξιοποιούν τη γεωγραφική τους θέση μεταξύ των αγορών και ε, ζωνών ορών, κάτι που τους ωφελεί. Εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό και όχι να μη μυρολατρικά να ψημυρούμε. Επίσης, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τεράστιες υπεκφυγές, κολλησιεργία για την ε, χωρητικότητα των αεροδρομίων, τη δημιουργία νέων διαδρόμων. Η αεροπορία αντιμετωπίζεται ως αγελάδα προσάρμαγμα. Και ε, έχουμε πολλά τέλη, έχουμε τα πρώην καλύτερα αεροδρόμια, τα πιο επικερδή και έξι από τα δέκα παγκοσμίως επικερδή είναι στην Ευρώπη. Αλλά τα, οι φόροι, τα τέλη αεροδρομίου επιβαρύνουν κυρίως τις αεροπορικές εταιρείες γιατί τα τέλη είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων στα δικά μας αεροδρόμια. Δηλαδή οι κυβερνήσεις λένε ότι δικαίωμά μας είναι. Αλλά δεν μπορείτε να απαιτείτε από άλλες κυβερνήσεις να υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση. Θα πρέπει να μάθουμε από τις δικές προσεγγίσεις και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πώς μπορούμε τώρα να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Άλλο ανταγωνιστικότητα, άλλο ανταγωνισμός. Παρόλο που μερικές φορές κατά λάθο και εσφαλμένα το συνώνυμα. Ε, μόνοι μας έχουμε επιβάλει ε, φραγμούς ενιαίοι ευρωπαϊκοί εθέρες. Σίγουρα χρειάζονται. Εδώ και 10 χρόνια το συζητούμε, αλλά δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο. Έχουμε κατακαιρματισμένο ένα αέριο χώρο. Μας κοστίζει 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επίση, έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εμπορία εκπομπών. Εμεί ταχθήκαμε υπέρ του συστήματο ε, εμπορία εκπομπών, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν ε, περιβαλλοντικά υποφελές, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προτιμούμε τώρα μια παγκόσμια λύση, ώστε το ευρωπαϊκό ETS να γίνει περιττό. Δεν μπορούμε όμω να έχουμε ε, διπλές επιβαρύνσει ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να πληρώνουν και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ETS, έχοντας πολύ περισσότερο βάρος και τέλη να καταβάλουν. Τώρα, πιστεύουμε στην φιλελευθερωποίηση, αλλά δεν έχουν απελευθερωθεί όλοι οι τομεί δυστυχώ. Έχουμε όλο και περισσότερες ευκαιρίες χάρη στην απελευθέρωση και η σύμβαση του Σικάγο δίνει έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών. Νομίζω ότι αυτό είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξασφαλίσει ισότητα, ίσες ευκαιρίες για όλες τις αεροπορικές εταιρείες, για να έχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Από εσά εξαρτάται ε, να εξασφαλίσετε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και εμεί να είμαστε εύρωστοι και να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις υπόλοιπε εταιρείε. Και όταν έχουμε απελευθερωμένε συμφωνίες όπως με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, ταυτόχρονα διαφυλάσσουμε σε πολλές περιπτώσεις ε, κάποιες θέσεις εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιριών οι αμερικανικές εταιρείε είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Επίσης δεν απελευθερώθηκε η ιδιοκτησία και ο έλεγχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχώς ε, ε, ε οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν τη Fly America, μια εξαιρετικά προστατευτική πολιτική. Και μάλιστα η Αμερική που πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση των αγορών εξακολουθεί να επιβάλλει ιδιαίτερα προστατευτικές διατάξεις και πολλοί παραπονιούνται για τις πολιτικές και των χωρών του, του κόλπου. Αλλά νομίζω ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και σταθμά πολλές φορές στις προσεγγίσεις μας. Η τεχνολογία με εμποδίζει εδώ να προχωρήσω. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να συνεχίσουμε στο δρόμο της απελευθέρωσης. Μόνο έτσι θα πρέπει να προωθήσουμε την εντολή που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Συμβούλιο και να διεκδικήσουμε τις ευκαιρίες για τις αεροπορικές εταιρείες. Και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να ετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στον υψηλό ανταγωνισμό. Και ο κανονισμός 868 μας αποσπά την προσοχή γιατί επιβραδύνει τη διαδικασία των, της διαπραγμάτευσης των νέων εντολών και δημιουργεί συνθήκες δύσκολες. Και ακόμη και αν ευοδοθεί η διαπραγμάτευση με τον 868 δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες συνθήκες. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να παραμείνουμε στα χρονικά όρια. Οι αεροπορικέ εταιρείε ε, μπορεί να, είναι, να καθυστερούν πολλέ φορέ τι ε, προσγειώσει του. Ο κύριος Πόλατσεκ είναι ο επόμενο, ο οποίο είναι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Πιλότων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, μετά από τι παρουσιάσει αποφάσισα σε ισχυρό αποφάσισα να μην χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνολογία. Πρώτα απ' όλα θα σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μα δίνετε από την πλευρά τη Ένωση των Πιλότων για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντική ευκαιρία για μας. Να ξεκινήσω την ομιλία μου με μία παράθεση. Το στρατηγικό πακέτο αεροπορίας είναι μια, ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κλάδος αερομεταφορών ως συμβολέα στην ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τον τομέα μας, τον κλάδο μας. Ένα μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Δυστυχώς αυτή η παράθεση δεν ήρθε από την Ευρώπη αλλά από τις τρεις μεγάλες εταιρείες του Περσικού κόλπου. Γιατί εμείς λοιπόν ε, δεν ακολουθούμε αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνουμε τη σημαντική στρατηγική σημασία της αεροπορίας, αλλά όχι τόσο καλά όσο οι χώρες του Πεσκού κόλπου. Οδηγεί σε ανάπτυξη της εργασίας και συνδεσιμότητα, όπως ελέγχει, και συνδέει τις εξαγωγικές εταιρείε της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ανισομέρεια στην αγορά <clears throat> αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Υπήρου, σε βάρος των αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία πρώτα απ' όλα οι εταιρείε του Περσικού κόλπου έχουν αυξήσει την ικανότητα μεταφοράς τους προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 112%, οι ευρωπαϊκές εταιρείε έχουν μειώσει κατά 14%. Επίσης, έχουμε 250 αεροσκάφη μεγάλης αποστάσεως. Οι τρεις εταιρείε μοναχά, η Κατάρ, η Etihad και Emirates έχουν 604 αεροπλάνα που έχουν ε, παραγγείλει για μακρές διαδρομές. Τρεις φορές περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς. Τρίτον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία αύξηση για χωρητικότητα μεγάλων αποστάσεων. Πέντε φορές μεγαλύτερη ικανότητα έχουν οι εταιρείε του Περσικού κόλπου έναντι του 2005. Τέλος, η λειτουργία ενός ε, αεροπλάνου ε, ευρέως ε, μεγάλου εύρους δημιουργεί περίπου 500 θέσει εργασία στον ε, Περσικό κόλπο η λειτουργία ενός τέτοιου αεροπλάνου θα οδηγήσει μονάχα σε 50 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Επομένως, η απώλεια οδηγήσε, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή ο ευρωπαϊκός κλάδος θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε συνθήκες ανταγωνισμού με τις άλλες εταιρείε, αλλά χρειαζόμαστε ή σε συνθήκες ανταγωνισμού. Γιατί κάναμε όλες αυτές τις προσπάθειες για να απαγορεύσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και να φιλελευθερωποιήσουμε την αγορά μας, άμα τώρα δίνουμε τον έλεγχο της αγοράς μας σε εθνικά επιδοτούμενες εταιρείε όπως αυτές του Περσικού Κόλπου. Γιατί ο ανταγωνισμός με άλλες περιοχές του κόσμου όπως παραδείγματος χάρη με τις χώρες ΑΣΕΑΝ δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενος. Οι άμεσες συνδέσεις μεταξύ των δύο αυτών τμήματων του κόσμου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω του ανταγωνισμού από τις ε, αεροπορικές εταιρείε του Πεσκού κόλπου που ουσιαστικά αντικαθιστούν και υποκαθιστούν τις ευρωπαϊκές πτήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι η διπυρωτική μας συνδεσιμότητα υποφέρει πάρα πολύ και επίσης ε, το θέμα του αν θα πρέπει να επιτρέψουμε επενδύσεις από τις χώρες του Περσικού κόλπου στις αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης. Έχουμε δει ότι αυτές οι επενδύσεις δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη συνδετιμότητα ή ανάπτυξη, αλλά απλώς διατηρούν υπερβολική ικανότητα μεταφορά σε μια ε, κορεσμένη αγορά και οδηγούν και σε απώλεια θέσεων απασχόλησης. Αυτές οι επενδύσεις σημαίνουν ότι η άμεση συνδεσιμότητα μειώνεται και αντικαθίσταται από έμεσε συνδέσει μέσω των χωρών του Περσικού κόλπου. Οι συνέπειε για την οικονομία μα αρχίζουν να γίνονται ορατέ όπω είπα προηγουμένω, χρειαζόμαστε ίσε συνθήκε ανταγωνισμού για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τι μεταφορικέ εταιρείε τρίτων χωρών. Αυτό πώ θα γίνει όμω, Χρειάζεται καταρχήν πρόσβαση στην αγορά. Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αγορά, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων θέλουν να ταξιδέψουν και πολλοί από αυτούς θέλουν να κινηθούν μέσα στην Ευρώπη και περισσότεροι. Αλλά αυτή η πρόσβαση στην αγορά μπορεί να ε, ανταλλαγεί μόνο μια φορά με αντίστοιχες παραχώρησεις. Για να μπορούμε να έχουμε λοιπόν τη σωστή ανταγωνιστικότητα και η Κομισιόν να έχει τη σωστή συμφωνία με τις χώρες του Πεσκού Κόλπου θέλουμε αυτές τις συμφωνίες να είναι αυτό που πρέπει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική εντολή που να βασίζεται σε ίσο ανταγωνισμό, ενώ πρέπει να διατηρηθούν τα δικαιώματα για πτήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για να εξασφαλίσουμε σαφή, ε, σαφείς ρήτρες για τις κρατικές επιδοτήσεις των περιβάλλον, την ανθρώπινη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Χρειαζόμαστε να υπάρχει και μια εύρωστη κοινωνική ρήτρα. Πρωτού προχωρήσουμε θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα τι κερδίζουν οι Ευρωπαίοι από τέτοιες συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και ότι θα έχουμε καλύτερα εργαλεία αμυντικού χαρακτήρα όπως η Οδηγία 868 του 2014 για τις ε, <clears throat> επιδοτήσεις καταχρηστικές από τρίτες χώρες. Αυτό όμως δεν είναι τμήμα του πακέτου αεροπορίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει σύντομα μια νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν. Τέλος, ό,τι αφορά την επένδυση από εταιρείε του Περσικού κόλπου, ίσως αυτή είναι απλώς δούρη ήπη οι πτάμενοι βέβαια, οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ευρώπη έχει μια πάρα πολύ φιλελεύθερη πολιτική για την ξένη διοξία των εταιριών τους. Αυτό μόνο σε διμερή βάση θα μπορούσε να λειτουργεί. Θα πρέπει να ενισχύουν αυτοί οι κανόνε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο έλεγχο των ευρωπαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκά χέρια και όχι σε ξένα χέρια. Ε, έχω ξεπεράσει τον χρόνο μου, λοιπόν κυρίε και κύριοι, σταματώ εδώ. Ένα πράγμα είναι σαφέ δεν μπορεί κανένα κλάδο να, υποστη... να ανταγωνιστεί χωρί τι ίσε συνθήκε ανταγωνισμού και θέλουμε την υποστήριξή σα. Well. And... Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριο Ολιβιέ Γιάνκοβιτ, που είναι Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Έχω μία παρουσίαση να σας κάνω ε, βασίζομαι στην ε, κοινοβουλευτική βοήθεια για να προχωρήσω τις διαφάνειες. Ε, επόμενη παρακαλώ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αποδίδουν μεγάλη σημασία στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων, διότι έτσι αυξάνουν τις προορισμούς τους οποίους εξυπηρετούν για τους επιβάτες και για τα φορτία και αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και πυρήνα ε, ε, των επιχειρήσεών μα, ε, Μεγιστοποίηση παραγωγικότητα για τους καταναλωτές αλλά και η στήριξη των θέσεων. Είμαστε υπέρ λοιπόν φυσικά του ανταγωνισμού και πιστεύουμε πως ο ανταγωνισμός θα έπρεπε καταρχάς να επιτρέπει να οδηγούμεθα σε περισσότερες διασυνδέσεις, περισσότερη κατανάλωση και περισσότερα επιχειρησιακά ωφέλη. Και αυτό έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που δημιουργήσε την εσωτερική αγορά για την αεροπλοεία που βασίστηκε στην ε, αρχή των ανοιχτών ε, εθέρων ε, και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τα ωφέλη που για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα όμως έχουμε νέα εστίαση, εξωτερική διάσταση, πώς μπορούμε να κινηθούμε πέρα από την εσωτερική μας αγορά ως Ευρώπη. Η εξωτερική διάσταση είναι πολύ σχετική για την αεροπλοή, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε με παγκόσμια μετακίνηση του, της παγκόσμιας οικονομίας σταδιακά προς τις αναδυόμενες αγορές. Αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη όλα είναι και περισσότερο εξαρτάται από το εξωτερικό εμπόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι στο πλαίσιο αυτό οι διασυνδέσεις και η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στις αναδυόμενες αυτές αγορές είναι στρατηγική σημασίας για την Ευρώπη τη σήμερα ημέρα. Αυτό που είδαμε είναι ότι βεβαίως αυτό συνοδεύεται από νέες ε, δυνάμεις και νέες αεροπορικές εταιρείε με πολύ, μεγάλες, ε, ε, πολύ μεγάλη ισχύ. Επηρεάζουν αυτό, αυτές την αγορά, αλλά όχι όπως το παρελθόν οι, αγορές, οι αεροπορικές εταιρείε χαμηλού κόστους. Όσον αφορά την στρατηγική σημασία λοιπόν της, των διασυνδέσεών μας, ε, ε, θα πω ότι είναι σαφές πως οι διασυνδέσεις σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη. 10% ανάπτυξη στις ε, αεροπορικές διασυνδέσεις οδηγεί σε συν 0,5% στο ΕΠ και φυσικά αυτό δεν θέλει να το χάσει η Ευρώπη. Πολλή συζήτηση γίνεται για το ίσους όρους ε, του παιχνιδιού και τίνω να συμφωνώ με τον ΩΣΑ ότι πρόκειται για παραπλανητική έννοια η οποία δεν έχει και μεγάλη σημασία στο τέλος για αυτά που συζητάμε σήμερα. Και γιατί, διότι ε, ίσοι όροι παιχνιδιού είναι πάντα άνηση. Ποτέ δεν πρόκειται να υπάρχει απόλυτα τέλειο, ε, τέλεια ισότητα και ούτε καν και είναι επιθυμητό αυτό. Γιατί, καταρχάς, λόγω της γεωγραφικής θέσης της κάθε χώρας, αν εστιάσουμε στις μεταφορείς του Περσικού κόλπου και βλέπετε πόσο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια οι δικέ του αεροπορικές συνδέσεις έχουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της γεωγραφικής τους θέσης που τους επιτρέπει να φτιάχνουν ε, ε, ε, διαδρομές ε, τις οποίες ε, εποφελούνται από πολλές οικονομικές απόψεις για τα αεροσκάφη τους. Ε, επίσης, ε, εξαρτάται ε, το ίση όρια από τις εθνικές πολιτικές. Δημόσια χρηματοδότηση είναι εκτεταμένη εκτός Ευρώπης και στη ΣΥΠΑ. Ασφάλεια στη χρηματοδότηση και πάλι η Ευρώπη εδώ είναι μοναχικός καβαλάρης και ζητά από τη βιομηχανία της να πληρώσει για την ασφάλεια στην αεροπλοεία. Και για τη φορολογική πολιτική είναι η μόνη που η Ευρωπαϊκή Ένωση που φορολογεί την αεροπλοεία. Αυτές οι επιλογές είναι θεμητές επιλογές όταν κανείς αποφασίζει πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία του. Και θα πρέπει τέλος έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία για τις σώτιμου όρου ανταγωνισμού. Έχουμε καταρχήν εγκάρσια ολοκλήρωση μεταξύ των αεροδρομίων και των εθνικών αερογραμμών και πλήρω ολοκληρωμένο μοντέλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά έχουμε και ε, ενδιάμεσα μοντέλα μη ολοκληρωμένα, όπως αυτό που ισχύει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί τα αεροδρόμια είναι δημόσια αγαθά και ανήκουν στο δημόσιο. Ε, επίσης, ε, Ποια είναι τα κέρια στοιχεία της νέας πολιτικής αεροπορίας. Εδώ βλέπετε μια φράση που την πήρα από την ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Ντουμπάι. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την πορεία της ε, ιστορίας της, ε, της αεροπορίας και να ε, βελτιώσουμε την ευημερία και την συνολική κατάσταση του Ντουμπάι. Αυτό, αυτό είναι ένα σημαντικό όραμα και χαιρόμαστε που το πακέτο για την αεροπορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Από αυτήν την άποψη η αναζήτηση του ισότιμου ανταγωνισμού είναι μάλλον ε, ουτοπία, φαντασίωση. Και πολύ συχνά είναι μια συγκαλυμμένη προσπάθεια προστατευτισμού. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ανοιχτή εθέρε και ισότιμος δίκαιος, θεμητός ανταγωνισμός. Και τι εννοούμε όταν λέμε θεμητό ανταγωνισμό, όπως είπε και ο κύριος από τον ΩΣΑ, θέλουμε ισότητα ευκαιριών, όχι ισότητα αποτελέσματος, ε, δηλαδή εξορρόπηση αποτελεσμάτων των αερογραμμών. Τώρα, ποια είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πάμε στην επόμενη ε, διαφάνεια. Οι διμερείς ε, συμφωνίες και η ρήτρα της, της κοινότητας δεν είναι η λύση γιατί η διμερής ε, προσέγγιση δημιουργεί πρόσκομα στον ανταγωνισμό. Δεν εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση και δυστυχώς εξωθεί τα αεροδρόμια ε, εκτός του ανταγωνισμού και της ε, διαβούλευσης. Δεν είναι σωστή η ρήτρα επίσης για την κοινότητα, γιατί δεν οδηγεί σε ομοιόμορφη ερμηνεία. Ούτε προωθεί την ευρωπαϊκή αεροπορία. Θέλουμε λοιπόν συνολικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα στηρίζονται σε ανοιχτού εθέρε, που είναι απαραίτητη προπόθεση για το θεμητό ανταγωνισμό. Επίση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό το θεμητό ανταγωνισμό και να τον ελέγξουμε. Γιατί πολλά συζητώνται για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ρήτρα ανταγωνισμού στι συμφωνίε αυτέ. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οικουμενική αυτή η ρήτρα, να, να ε, αντιμετωπίζει όλους και τους εξωκοινωτικούς με τον ίδιο τρόπο, να μην προβλέπει διακρίσεις, να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις των ξένων αεροπορικών εταιριών, ε, συμφωνίες για συγκεκριμένα θέματα κατά της συγκέντρωσης, συμφωνημένες διαδικασίες για τις διαφορές και Τέλος, πέραν της ε, ρήτρα ε, θεμετού ανταγωνισμού, χρειαζόμαστε μια πιο ρεαλιστική και σφαιρική προσέγγιση για την αεροπορία. Και από αυτήν την άποψη, το πακέτο αεροπορίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί το σωστό δρόμο. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την έλλειψη της, ε, του προβλήματος στη χωρητικότητα των αεροδρομίων. Πώς αντιμετωπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αεροπορία. Γιατί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογεί την αεροπλοεία. Έχουμε επίσης υψηλό κόστος ε, λόγω του των κανονιστικών ρυθμίσεων και περιορίζουμε και τις δημόσιες δαπάνες. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, αυτό που είπε ο Τζον για τα τέλη αεροδρομίου. Τα αεροδρόμια ουσιαστικά ενισχύουν ε, τις αεροπορικές γραμμές που δεν πληρώνουν στο ολόκληρο το, το τέλος των αεροδρομίων γιατί από αυτή την άποψη ε, ξεκονομούν ε, κάποια στοιχεία. Και η όλη η ρητορική για το, τέλ, για το τέλος των αεροδρομίων ουσιαστικά προσπαθεί να, δικαιολογήσει την ανικανότητα κάποιων, αεροπορικών εταιριών στον ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της στρατηγικής αεροπορίας. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της διεθνούς του Διεθνού Οργανισμού Ασφάλεια τη Αεροπλοεία. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι εντολέ και ελπίζουμε και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό να δώσει την εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεκινήσουμε τι διαδικασίε και την... το έτο. Σα ευχαριστώ και τον τελευταίο ομιλητή τον κύριο Κλάου Γκάιλ, επικεφαλή τομέα στην DigiMove για τον τομέα τη εξωτερικού αεροπορικού κλάδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ. Το <clears throat> αντικείμενο που έχετε επιλέξει είναι πολύ ενδιαφέρον και τα ερωτήματά σας είναι ιδιαίτερα εύστοχα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω τα ερωτήματα αυτά. Και να απαντήσω και στα ερωτήματα μπορεί να έχουν τα έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ξεπεράσω και το χρόνο μου αλλά είναι και αυτό <clears throat> προ όφελο τη ισότητα ανταγωνισμού και η Κομισιόν. θα πρέπει να λιγάκι. Ο ανταγωνισμός <clears throat> στην διεθνή αεροπλοεία, η φιλελευθερωποίηση και το πώς θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε συμφωνίες και με ποιον αυτά είναι θέματα τα οποία αναμοχλεύουν τα πάθη στις συζητήσεις και είναι θυμήματα της στρατηγικής αεροπορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεκρίθησαν στις 7 ε, Σεπτεμβρίου και η Επίτροπος κυρία Μπούλτς ήρθε ενώπιον της Επιτροπής σας να παρουσιάσει τη συζήτηση αυτή για τη φιλελευθερωποίηση στον αεροπορικό κλάδο. Υπάρχει ένα παράδοξο μερικές φορές. Παρουσιάζεται η Ευρώπη ως προστατευτική και περιοριστική σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πιο φιλελευθερωποιημένο και ανοιχτό κλάδο αεροπορία στον κόσμο και αυτό ήταν μια μεγάλη πτυχία και έχει τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο πετάμε προ όφελο των πολιτών μα. Δίνει και νέε ευκαιρίε για τι επιχειρήσει μα. Η εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα φιλελευθερωποιηθεί πλήρω εδώ και 20 χρόνια και έχουμε ξεχάσει πω επετέφθη κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά όμως τον αντίκτυπο που οδήγησε σε περισσότερο ανταγωνισμό, νέες διαδρομές, μεγαλύτερη ε, συνδεσιμότητα, μεγαλύτερη κινητικότητα για τους ανθρώπους, όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Οι εταιρείε χαμηλού κόστους, που είναι τα παιδιά ουσιαστικά των μεταρρυθμίσεων αυτών και της έχουν το 50% της ε, αεροπορικής κίνησης και μεγαλώνουν ακόμα. Η Ενέ είναι ο μεγαλύτερο αερομεταφορέα σε ό,τι αφορά τον αριθμό επιβατών, φτάνει τα 5 εκατομμύρια φέτο. Έχουμε φιλεδοποίηση τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πια εθνικέ εταιρείε, αλλά ευρωπαϊκέ εταιρείε και ομίλου εταιριών επί τη βάση κανόνων αδειοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πιο φιλελεύθερους κανόνες για ξένες επενδύσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείε από τι άλλες περιοχές του κόσμου και είδαμε πολλές επενδύσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείε, όχι μόνο από τον Περσικό κόλπο όπως είπαμε. <clears throat> Αλλά φυσικά απαιτούμε από τους ξένους επενδυτές να συμμορφώνονται με τους κανόνες μας. Ένα από τα κέρια διδάγματα που έχουμε αποκομίσει από την ανάπτυξη του εσωτερικού κλάδο αεροπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όσο πιο φιλελευθερωποιούμε τον κανόνα, τόσο πιο απαραίτητο είναι να έχουμε κάποιου κοινού κανόνε Αυτό αφορά όχι μόνο την αεροπορία, αλλά όλους τους οικονομικούς τομείς της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης τεχνικών προτύπων κοινών κανόνων που να ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στεναρής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για τις κρατικέ επιδοτήσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ στεγατές εξουσίες για να τα εξασφαλίσει όλα αυτά. Μόλον τούτο, ένα <clears throat> πλήρες, η πλήρης ισότητα ανταγωνισμού είναι μια φενάκι. Όλες οι εταιρείε έχουν τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχουν διαφορετικά πρότυπα, τα οποία εν τούτης ποικίλουν σε όλο τον κόσμο και μεταξύ εμπονωμένων χωρών. Πιστεύουμε βάσει της εμπειρίας μας με την εσωτερική αγορά ότι οι ανοιχτές αγορές είναι ο καλύτερος χώρος για την διεθνή αεροπορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια έχει υπογράψει φιλόδοξε και πλήρε συμφωνίε αεροπορικού χαρακτήρα με τον Καναδά, τι ΗΠΑ, το Μαρόκο, τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, την Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ και υπάρχει και μια επικείμενη συμφωνία για το θέμα του Γιβραλτάρ και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τινησία και την Βραζιλία. Ελπίζουμε να περατώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τη Βραζιλία στην αρχή του επόμενου χρόνου. Αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των συμφωνιών είναι μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, ενισχυμένη συνεργασία από όλες τις πτυχές της αεροπορίας και το σωστό πλαίσιο ανταγωνισμού μέσω σύγκλησης στα αριθμιστικά θέματα τα αποτελέσματα με την αύξηση της κίνησης είναι απτά. Οι περισσότερες χώρες έχουν αναφέρει ότι έχει διπλασιαστεί η κίνηση. Οι πτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής και Δυτικών Βαλκανίων έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου έχουν υπερδιπλασιαστεί από 5,6 επιβάτες σε 12 εκατομμύρια. Το 2012 υπολογίσαμε ότι τότε ήδη η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και το Μαρόκο που έγινε το 2006 είχαν οδηγήσει σε ένα πλεόνασμα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές και μείωσαν τις, τους ναύλους κατά 40%. Αλλά και εδώ και πάλι σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά θέματα πιστεύουμε ότι όσο πιο φιλελευθερωποιημένες και παγκοσμιοποιημένες είναι οι αγορές τόσο πιο ε, εν τούτης, ε, απαραίτητο είναι να υπάρξουν κοινοί κανόνε στο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απρόοπτο στον διεθνή χώρο. Ακούσαμε και από άλλου ομιλητέ να λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα παγκόσμιο νομικό πλαίσιο στον ΠΟΕ, παραδείγματο χάρη, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ΠΟΕ έχει καθορίσει ένα αριθμό κανόνων για το τι είναι οι επιδοτήσεις, ποιες επιδοτήσεις απαγορεύονται, πώς μπορεί κανείς να λάβει αντίμετρα εναντίον των ε, επιδοτήσεων. Για κάποιο λόγο όμως ο αεροπορικός κλάδος δεν καλύπτεται από τους κανόνες του ΠΟΕ και οι κανόνες του ΙΚΑΟ δεν δίνουν κάποιες παγκόσμιες δεσμευτικές νομικά ρυθμίσεις για την, τον αεροπορικό κλάδο, γιατί η ΚΑΟ ασχολείται περισσότερο με τα θέματα τα τεχνικά και της ασφάλειας. Και δεν υπάρχουν και τέτοιοι κανόνες συνήθως στις διμερείς συμφωνίες που διέπουν τη μεγαλύτερη περίπτωση μέρο των αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο. Δεν θα βρείτε ρήτρε και πρόνοιες σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά υπεριφαλλοντικά στοιχεία ή τον ίσο ανταγωνισμό στι διμερεί αυτέ συμφωνίε που έχουν κάνει οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Αυτέ οι διμερεί συμφωνίε αφορούν κυρίω την πρόσβαση στην αγορά και κυρίω του περιορισμού στην πρόσβαση τη αγορά. Απουσία εν τούτη ενό τέτοιου πλαισίου, απουσία κανόνων σε διμερεί συμφωνίε του προ την κατεύθυνση αυτή, είναι θεμητό και δίκαιο για την Ευρώπη να πάρει ένα ηγετικό ρόλο, να προτείνει κανόνες, να αναπτύξει εργαλεία για να εξασφαλίσει τον ανοιχτό και ελεύθερο ανταγωνισμό σε ένα κλάδο που είναι όλο και πιο παγκοσμιοποιημένος και επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειες για συμφωνίες αεροπορικού χαρακτήρα που να βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Αυτό πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 στην ανακοίνωση για την εξωτερική πολιτική αεροπορία. Και τώρα έχουμε νέα στρατηγική για την Ευρώπη ε, που μάλιστα τη στήριξε και η Επιτροπή σας και συσσωμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείναμε ένα φιλόδοξο πακέτο εντολών και δεν θα επαναλάβω εδώ αυτά που είπα προηγουμένως για τις ε, χώρες της επιμέρους. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα θέλετε. Πάντως το πακέτο μας είναι φιλόδοξο για διαπραγμάτευση πανευρωπαϊκών συμφωνιών και μάλιστα βασική προτεραιότητα της ε, εξωτερικής μας πολιτικής για την αεροπορία είναι να μπορέσει ο τομέας της ευρωπαϊκής αεροπορίας ε, να διεισδύσει σε αναδυόμενες ε, αγορές και οικονομίες και μέσω ενοχικών σχέσεων με τους εταίρους μας να προβλέψουμε ένα προβλέψιμο νομικό περιβάλλον για να εμβαθύνουμε τις αεροπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Μήπως θα μπορούσατε να βάλετε τελεία κύριε Γκάιλ. Θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών με τις χώρες του Περσικού κόλπου, για παράδειγμα, προσφέρουν την καλύτερη δυνατή και περιεκτική βάση για να γεφυρώσουμε τις ανησυχίες και να ε, ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες ε, αφωτέρων των πλευρών. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι στη διαπραγματεύση και συμφωνίες ε, να δημιουργήσουν ωφέλη και ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές και κυρίως να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο που να ενισχύει ε, την αγορά, την πρόοδό της, ε, το άνοιγμα της αγοράς και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό και μάλιστα είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να πάει χαμένη. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και περιμένουμε ε, την εντολή από το Συμβούλιο, από την Ολλανδική Προεδρία, ώστε να ξεκινήσουμε σοβαρά και τις, δύο τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες αυτές. Ο θε... βέβαια, η ισότιμος ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε προστατευτισμό ούτε να υποκαταστήσει τις ε, προσπάθειες που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο κλάδος της αεροπορίας για να παραμείνει ανταγωνιστικός και τα μέσα για διαφύλαξη του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά, αλλά είναι το ίστατο μέτρο σε περίπτωση που τεκμηριώνονται επιζήμιες ή αθέμετες πρακτικές. Και μάλιστα ε, η αναθεώρηση του κανονισμού 868 που θα λάβει χώρα το 2016 ε, θα πρέπει ε, να αποτρέψει να θέμει τον ανταγωνισμό και όχι να εμποδίσει το θεμητό ανταγωνισμό. Θέλουμε να στηρίξουμε τον ανταγωνισμό και αυτό από τα κράτη-μέλη, τι αεροπορικέ εταιρείε, τα συμβαλόμενα μέρη, του ενδιαφερομένου και τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα. Λυπούμε που μακρηγόρησα και υπερεύει το χρόνο, γιατί έτσι πραγματικά εγώ δημιούργησα συνθήκε άνισου ανταγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή σα Μεταφορών και Τουρισμού για την αμέριστη υποστήριξη και την αδιάλειπτη βοήθειά σα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην αεροπορία και στις προτινόμενες από εμάς εντολές όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τον ανοιχτό και θεμητό ανταγωνισμό προς όφελος και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Φυσικά, όπου τέτοια μέτρα είναι δικαιολογημένα και απαραίτητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, ε, μιλήσατε το διπλάσιο χρόνο από αυτό που σας είχαμε δώσει. Τώρα ολοκληρώθηκαν ε, οι παρουσιάσεις, οι εισηγήσει και τώρα έχουμε λίγο χρόνο για να θέσετε ερωτήσεις και για να απαντήσετε εσείς ως ειδικοί. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές, τους τρεις εισηγητές σε μια ωρίτσα πήραμε μια εικόνα, καλή εικόνα. Α, πόσο χρόνο έχω πρόεδρε, γιατί δεν μου είπατε για να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα. Α, λίγη. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν, Πρόεδρε, ότι ε, θέλω... πήραμε μια καλή εικόνα για το τι έχουμε ακόμα να κάνουμε. Χαίρομαι που Υπάρχει αυτό το πακέτο για την αεροπλοεία, το περιμέναμε εδώ και καιρό. Τουλάχιστον τώρα έχουμε ένα έγγραφο που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσεις, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Στο όνομα του Ευρωκοινοβουλίου πιστεύω ότι ε, θα θέλαμε το ίδιο και για τι ε, οδικές μεταφορές αλλά και για τις θαλάσσιες μεταφορές και ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω. Τρει κατευθυντήριες γραμμές, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεύτερον, ο ανταγωνισμό ε, υπάρχει και είναι αθέμετος. Και τρίτη κατευθυντήρια γραμμή. Εμείς στην Ευρώπη τα κάνουμε καλύτερα. Πρώτη διαπίστωση, ναι, ο κόσμος έχει αλλάξει, αλήθεια είναι αυτό. Βλέπουμε ότι το κέντρο βαρύτητας περνά από τη Δύση στην Ανατολή και δεν μπορούμε να αρκούμεθα και να διαμαρτυρόμαστε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμό. Αυτό έχει ήδη γίνει, είναι ένα γεγονός, πρέπει εμείς αυτό να ανταποκριθούμε. Οι ασιατικές χώρε είναι σε πλήρη άνθηση και η Ευρώπη πρέπει να μπορέσει να να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεύτερη διαπίστωση, δεν είμαστε τόσο μικροί. Επανειλημμένως ε, μας είπατε ότι ο ΙΚΑΟ πρέπει να πάρει την σκητάλη. Εγώ, Πρόεδρε, απογοητεύομαι όταν βλέπω την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί ο ΙΚΑΟ, ενώ άλλοι προχωρούν με βήματα ταχύ. Κύριε Λαμπρόζο, πώς μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με την ταχύτητα των εξελίξεων παγκοσμίω. Δεύτερη ερώτηση, η όροι του παιχνιδιού. Ποτέ είπατε δεν ίσχυει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά στις κάτω χώρες μιλάμε για το ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε και η, η του χωριού. Ε, όταν ε, ακούμε να λέει ο κύριος Λαμπρόζο τέτοια, νιώθουμε σαν να είμαστε ο χαζός του, του, του χωριού, τα κορόιδα και ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μια χαρά τη δουλίτσα τους. Όχι. Αν οι υπόλοιποι δεν είναι ε, έτοιμοι να ανοίξουν τη συζήτηση, να ανοίξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, τότε ούτε και εμείς και να πούμε και εμείς δεν αλλάζουμε τις νομοθεσίες μας και ό,τι γίνει έγινε μετά. Σώσανε αυτό σωθεί το, αλλά όχι, δεν θέλουμε εμεί κάτι τέτοιο. Μήπως υπάρχουν υπερβολικά πολλές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη. Δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας και εδώ μιλώ για τα πληρώματα δεν κοστίζει πάρα πολύ. Οι θέσεις απασχόλησης δεν κοστίζουν υπερβολικά πολύ. Και τρίτον, απελευθέρωση μπορούμε να απελευθερώνουμε, αλλά πρέπει όλοι να τα κάνουν αυτό το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, εμείς να απελευθερώνουμε. Δεν αρκεί να ανοίγουμε εμείς τις πόρτες μας. Και τέλος, Πρόεδρε, τα κάτι μελη Αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δεχτούν το πακέτο για τους ανοιχτούς ευθέρες ή το ΣΕΖΑΡ. Τι να κάνουμε τώρα. Απευθύνω αυτή την έκκληση στα κάτι μέλη. Ε, ανοίξτε το πακέτο για την αεροπλοεία. Οι Ισπανοί μόλις έκαναν εκλογές. Και αν οι Ισπανοί λύσουν το θέμα τους, εμείς σε δύο μήνες στην Ολλανδική Προεδρία θα το λύσουμε όλο. Ευχαριστώ. Είπαμε τρία λεπτά για τους συντονιστές. Ο Ισμαήλ. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω μια οργανωτική αίτηση. Μήπως μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις ε, ε, παρουσιάσεις στην κεντρική οθόνη και όχι δεξιά και αριστερά γιατί παθαίνουμε νευροκαβαλίκευμα προσπαθώντας να καταλάβουμε τι γίνεται. Ωραία. Και τώρα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φάντερ που λέει ότι πρέπει να θέσουμε σε τάξη τα του οίκου μας. Ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τόσα ανοιχτά εργοτάξια που δεν τα έχουμε συμπληρώσει. Παρουσιάστηκε εδώ ένα παράδειγμα και από τους ομιλητές. για το θέμα των ε, ανοιχτών ευρωπαϊκών εθέρων που είναι ένα ανοιχτό γιαπί. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα αυτά. Και ο κύριος Πόλατσεκ μας ε, προειδοποίησε για το τι σημαίνει να έχουμε μια απόλυτα ανοιχτή και ε, φιλελεύθερη αντιμετώπιση, αν κατάλαβα καλά. Δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση στο να υπάρξει ελευθερία και ανοιχτό πλαίσιο. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε και κάποια κριτήρια. Και γι' αυτό το λόγο θέλω και εγώ να δω τι ακριβώς θα μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του 868 κάθος 2014 σε ό,τι αφορά την ισότητα ανταγωνισμού. Φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ισότητα 100%. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά <clears throat> να προσπαθήσουμε να κινηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, δηλαδή να κρατήσουμε και ανοιχτή την αγορά και την ελευθερία ανταγωνισμού χωρίς να αυτοκτονήσουμε ουσιαστικά για τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Ποιες είναι οι δικές σας επιθυμίες σας σε σχέση με τις χώρες του Περσικού κόλπου και τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες. Προς την Κομισιόν, ποιες είναι οι κύριες επιτυχίες που καλύπτονται από τις συμφωνίες με τα κράτη του Περσικού κόλπου και πώς μπορείτε να ενισχύσετε τις ευρωπαϊκές εταιρείες έναντι αυτών των συμφωνιών. <clears throat> Πιστεύω επίσης ότι οι οδηγίες ελέγχου και εποπτείας θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αλλά θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε τους ελέγχους σε ό,τι αφορά τις δικές μας αεροπορικές εταιρείες και νομίζω ότι μία από τις τελευταίες παρουσιάσεις έθεσαν το, ενώ, το ερώτημα του αν θα πρέπει να καθορίσουμε και πάλι να επαναθεωρήσουμε τα όρια των δημοσίων χρηματοδοτήσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Να έχουμε λοιπόν κανόνες για κρατικές επιδοτήσεις, που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε όπως ελέγχθη αυτό το, αυτή την ισότητα ανταγωνισμού. Και κατά τα άλλα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονό ότι η Κομισιό παρουσιάσει το πακέτο αεροπορικών θεμάτων. Η Γεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ από την πλευρά των φιλελευθέρων θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές σήμερα. Μια πρώτη παρατήρηση. Έχουμε ήδη το θέμα αυτό με το αεροπορικό πακέτο. Είναι απέτησή μας να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση της αεροπορίας στην Ευρώπη. Βλέπουμε πάρα πολλούς να θεωρούν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση συρρήκνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε εμείς να βελτιώσουμε τη θέση μας στον αεροπορικό κλάδο. Επίσης υπάρχουν στον αεροπορικό κλάδο πάρα πολλές θέσεις εργασίας, αεροπορικές εταιρείες, στα αεροδρόμια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας. Και επίσης και στην κατασκευή αεροσκαφών. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί γίνεται αυτή η εστίαση στις χώρες του Περσικού κόλπου Δεν μίλησε κανεί παραδείγματο χάρη για το αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη που έχει περίπου αντικαταστήσει ω κόμβο ε, αεροπορικών συνδέσεων την Φραγκφούρτη. Αυτές είναι οι πρώτες μου παρατηρήσεις και τώρα κάποια σχόλια κατευθείαν προς τους ομιλητές. Κύριε Λαμπρούσο, είπατε ότι δεν υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού, είναι μια ψευδέστηση. αν <clears throat> κατάλαβα, θέλετε να έχετε μια βασική σειρά ορισμών σε επίπεδο ΙΚΑΟ. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Η ΙΚΑΟ δουλεύει με χελωνοδρομικές διαδικασίες όπως είδαμε και στο ETS για τον κύριο Καν. Είπατε χρειαζόμαστε μια ρήτρα ίσου ανταγωνισμού στις ε, συμφωνίες διμερούς χαρακτήρα. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, με τι μορφή θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ρήτρα και τον κύριο Χένλον Και εγώ συμφωνώ μαζί σα. το ETS πρέπει να πάρει παγκόσμιο χαρακτήρα και όχι μονάχα ευρωπαϊκό. Είπατε το 868 ε, είναι μια διαδικασία που πρέπει να επιβραδυνθεί. Γιατί, με ποιο στόχο θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τον κύριο Πόλατσεκ είπατε και εσείς, ναι, η ισότητα ανταγωνισμού αυτό είναι απαραίτητο οι εταιρείε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αλλά πώ θα τον επιτύχουμε αυτόν τον ίσο ανταγωνισμό, με ποιο τρόπο. Και από τον κύριο Γιάνκοβιτ. Είπατε και εσεί πάλι ότι δεν υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού. Και το ερώτημα είναι αν μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά μέσα από συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών κλάδων. Να έχουμε συμφωνίες που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός για την Κομισιόν δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ θα ήθελα να πω απλώ ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών όταν τι εκτελεί η Κομισιόν. Μα εκεί λένε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω πως ελπίζω να μην παραμείνει ανδροκρατούμενη η αεροπορία. Και θα ήθελα να διεκδικήσω μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στην αεροπορία. Ήρθα τρέχοντα από την Επιτροπή Περιβάλλοντο για να παρακολουθήσω την ακρόαση και θα πρέπει επίση τρέχοντα να επιστρέψω στην Επιτροπή Περιβάλλοντο για τη συνέχεια της συνεδρίασης. Πρώτα απ' όλα όμως ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν αναφέρατε και μια καθαρή αεροπορία. Ε, πώς βλέπετε τα εναλλακτικά καύσιμα και στην αεροπορία για να έχουμε μια αεροπορία που δεν θα ρηπαίνει το περιβάλλον. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών καυσίμων. Έχετε παραδείγματα χρήσης τέτοιων εναλλακτικών καυσίμων για να έχουμε πιο καθαρή και φιλοπεριβαλλοντική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των πιλότων και του πληρώματος καμπίνας, είναι σημαντικό θέμα και αφορά την ασφάλεια όλων μας και των επιβατών και του πληρώματος. Έγιναν κάποιες συμφωνίες για την εκπαίδευση, τις οποίες όμως τις υπαγόρευσαν οι αεροπορικές εταιρείες και δεν νομίζω ότι ε, τα κριτήρια εξυπηρετούν ιδιαίτερα την ασφάλεια, παρά περισσότερο τα συμφέροντα των ε, αεροπορικών εταιριών. Ε, λυπούμε γιατί όπως σας είπα δεν θα ακούσω τις απαντήσεις. Πρέπει να επιστρέψω τρέχοντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και κυρίως ασφάλεια. Ευχαριστώ και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καρίνα Αντέλη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε έξι καλεσμένους και βλέπετε ότι τρεις ε, συντονίστρες της ομάδας ε, έχουμε ε, για να σχολιάσουν αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι και για τα θέματα αεροπορίας μπορούν και οι γυναίκες να έχουν γνώσεις και δεξιότητες. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική πρόκληση με 1,5 ε, βαθμό, μη υπέρβαση το, το, της του πλανήτη ε, του 1,5 βαθμού. Σημαντικός και δεσμευτικός στόχος και θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η αεροπορία. Ε, θα έχουμε μια παγκόσμια αγορά και θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα για τι εκπομπέ και μετά το 2020. Θα είναι πολύ σημαντικό να τι ελέγξουμε για να μην περβούμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου στην αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν και η αεροπορία να αυξήσει τι φιλοδοξίε του. γιατί αλλιώ άλλοι τομεί θα πρέπει να καλύψουν το έδαφο αυτή τη ε, χαλαρής ε, ή μικρή φιλοδοξία. Είναι δίκαιο άλλοι τομεί να αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο για τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή καυσερίων, αντί να πρέπει και η αεροπορία να αναλάβει και τις δικές ευθύνες. Ε, η φορολογία είναι σημαντικό εργαλείο. Ε, η φορολογία επί της κυροσύνης του καυσίμου της αεροπορίας ακόμη εξετάζεται. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας που έχει χαρα... χαντακώσει την αεροπορία. Αλλά η ζούγκα που κυκλοφορεί, ε, που ισχύει μάλλον, ε, και το κοινωνικό ντάμπινγκ των αεροπορικών ε, εταιριών που κακομεταχειρίζονται τους υπαλλήλους τους. Αυτή, αυτός ο αθέμετος ανταγωνισμός επηρεάζει τις τιμές, το μισθολογικό κόστος και το γεγονός ότι έχουμε low cost εταιρείε, αλλά και εταιρείε του περσικού κόλπου που υποφελούνται από υπέρογες κρατικές ενισχύσεις και ε, καθιστούν ανέφικτο οποιαδήποτε ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών. Οπότε δεν έχουμε αυστηρούς κανόνε για το χρόνο για την ασφάλεια των επιβατών, για τα εργασιακά δικαιώματα. Όλοι αυτοί οι κανόνε θα πρέπει να εξασφαλίσουν θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό 868, γιατί ακόμη και σήμερα δεν εφαρμόζεται. Πώς λοιπόν θα αναλάβετε και εσείς ε, το μερίδιο των ευθυνών σας ε, σε αυτή την προσπάθεια. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου έχει απομείνει χρόνος. Μου έχει απομείνει χρόνος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ερώτηση ως προς το κόστος. Γιατί πολλά μας είπατε για την ανάγκη ανταγωνιστικότητας. Ρίχνοντας όμως μια ματιά ε, το τζίρο σας και τα κέρδη σας, βλέπω ότι η αεροπορία έχει αρκετά κέρδη για το 2016. Βλέποντας όμως την ΙΑΤΑ που υπολογίζει ότι οι ευρωπαϊκές αερογραμμές ε, θα έχουν καθαρό κέρδος 8,5 ε, δισεκατομμύρια ε, δολάρια με μεγάλο κόστος ανά επιβάτη πολύ μεγαλύτερο το κέρδος των ευρωπαϊκών εταιριών. Είναι διπλάσιο σχεδόν από το αντίστοιχο κατακεφαλή κέρδος των ε, αεροπορικών εταιριών του Περσικού κόλπου. Οπότε από άποψη κέρδους είστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους ανταγωνιστές σας. Και τέλος, έχετε στοιχεία για την εξέλιξη των ε, επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο για τα τελευταία χρόνια. Ο Πέτερ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αληθεύει. ότι Αυτές οι απαντήσεις πολλές φορές τις ε, εκμεταλλεύονται και οι τοπικές αρχές σε σχέση με τα αεροδρόμια της περιοχής και χρησιμοποιούνται και οι φόροι για να επιδοτηθούν οι εταιρείε χαμηλού κόστους για να μπορούν να έχουν κερδοφορία. Έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Τα επίπεδα αποδοχών, ε, οι οι συνθήκε που δουλεύουν οι πιλότοι, όλα αυτά που οδηγούν σε μεγάλη περιπλοκή της ε, ιδιωτικής του ζωής. Μια τέτοια κατάσταση ανταγωνισμού είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε. Ο ανταγωνισμός έχει να κάνει με το πώς η φαντασία μπορεί κανείς να αναπτύξει που βάζει κανείς την ε, έδρα μια ε, εταιρείας. Ή οι λεγόμενες δημιουργικές λύσεις σε σχέση με τα πληρώματα και που είναι η έδρα τους και όχι το πραγματικό τους σπίτι. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν φαντασία που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες χαμηλού κόστους για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κερδοφορία. Και αυτές οι εταιρείε προσπαθούν ακριβώς να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Ανεξάρτητα από το τι σημαίνει αυτό για το προσωπικό. για τον εκπροσώπο των ε, εταιριών χαμηλού κόστους. Γιατί δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε με τις ίδιες συνθήκες όπως με τις άλλες εταιρείε. Γιατί οι εταιρείε χαμηλού κόστους θα πρέπει να έχουν ένα πλεονέκτημα που προέρχεται από αυτές τις εφάνταστες λύσεις, ενώ οι άλλες εταιρείε δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι το ερώτημα μου εσάς. Σας ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι συντονιστές. Δεν θα σας προσκαλέσω να απαντήσετε σε τρία λεπτά βέβαια ο καθένας και μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι ομιλητές και μπορείτε μετά να απαντήσετε και πάλι. Να κάνουμε λοιπόν αυτή την ενδιάμεση απάντηση. Θα είμαι αυστηρός με τον χρόνο ομιλίας, τρία λεπτά το μάξιμο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος αυτή τη φορά. Για να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα. Κύριε Βάντερ Κέμπ, πώς μπορούμε να έχουμε ισότητα μεταξύ Ευρώπης και άλλων περιοχών. Υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Παραδείγματος χάρη βλέπετε την ε, προνομιακή θέση ορισμένων αεροδρομίων έναντι των άλλων και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανεί. Και επίση υπάρχουν και οι επιλογέ σε επίπεδο πολιτική που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν και κάποιε επιπτώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπήρξαν κάποιε συνέπειε από τι επιλογέ μα. Ε, αν δεν είμαστε έτοιμοι αυτό να το κάνουμε, ίσως θα πρέπει να τις επανααναθεωρήσουμε. Λέτε ότι δεν, θα μας, δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν, δεν πρέπει να μας τα κορόιδα. Υπήρχε μια αεροπορική εταιρεία πριν από 20 χρόνια που κανείς δεν την ήθελε. Γιατί έφερε τους επιβάτες στον κόμβο της και τις στέλνανε μετά σε άλλα μέρη. Λέγανε «Α, ήταν η KLM». Και θεωρείται ότι αυτό <clears throat> οι άλλες εταιρείες είχαν μεγάλο πρόβλημα μαζί της. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι και άλλες εταιρείες ακολουθούν το ίδιο μοντέλο. Δεν σημαίνει ότι Προσπαθεί κάτι να πιάσει άλλους κορώνε, είναι θέμα συνδεσιμότητα. Δεν είναι θέμα λοιπόν τέτοιο. Τώρα το να θέσουμε τα του οίκου μα σε τάξη. Είχαμε πολλά παραδείγματα από τι εταιρείε χαμηλού κόστου στην ε, Ευρώπη και τον εκπρόσωπό τη σε ό,τι αφορά τι φορολογικέ, πολιτικέ και άλλε πολιτικέ. Και τελικά ο δαρβινισμός λέει ότι οι πιο ικανοί επιβιώνουν. Αν συνεχίσουμε να προστατεύουμε την αγορά, τότε δεν υπάρχει προσαρμογή των εταιριών, γιατί μπορούν να παραμένουν αντιδαρβηνικές στο δίνεκες. Για τους βασικούς ορισμούς του ΙΚΑ, πόσο γρήγορα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ο ΙΚΑΟ είναι ένας διευκολυντής. Είναι οι χώρες που εκπροσωπούνται. Αν συμφωνούσαν οι χώρες αυτές θα προχωρούσαν. Δεν νοικά όπου καθυστερεί είναι οι χώρες που έχουν τις αντιρρήσεις τους εξαρτάται από αυτές να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο ΙΚΑΟ είναι μονάχα ένα φόρουμ για τα καύσιμα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης νέων καυσίων, ιδίως βιοκαυσίων. Βλέπουμε εναλλακτικά βιοκαύσιμα τα οποία μπορούν να ε, αναμειγνύονται με την κυροζήνη που χρησιμοποιεί τώρα χωρίς να αλλάξει η τεχνολογία αυτή. Στην COP21 ε, υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τα αναλλακτικά κάψιμα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό τις επόμενες δεκαετίες και αυτό είναι ένα από τα πράγματα στα οποία βασίζονται οι εταιρείε για να μειωθούν οι εκπομπές τους. Θέλουν να υπάρξει μηδενική αύξηση της ε, εκπομπής διοικητήριου του άνθρακος μέχρι το 2025 και μείωση επέκεινα. Και τέλος το θέμα των ε, επιδοτήσεων θέτεται των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων. Πρέπει να υπάρξει όμως καθαρή ένα σαφής ορισμός του τι είναι μια επιδότηση και μετά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ο οποίος να είναι διάφανος για να επαληθεύονται. Αυτό σε εθνικό επίπεδο ή σε παγκοσμίο επίπεδο δεν υπάρχει. Κρίμα είναι. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα αυτά και έχουμε τα θέματα αυτά που είδατε από την Αμερικάνικη έκθεση και την απάντηση των ε, Εμμυράτων, της εταιρείας Emirates, μιλάνε για άλλα αντάλλων και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ο κύριος Καν. Εγώ θα <coughs> απαντήσω στην κύριο Βάντερ, στα Ολλανδικά αν μου το επιτρέπετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείε, πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείε μάλλον στην Ευρώπη. Πρέπει αυτό να αλλάξει, συμφωνούμε. Δεν έχει βρεθεί η ισορροπία. Βλέπω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το φροντίσουν τώρα. Οι συνθήκες εργασίας όσον αφορά τι αεροπορικές εταιρείε. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει το προσωπικό τους, έχουν μειώσει δηλαδή το εσωτερικό κόστος τους. Όντως πρέπει να θίξουμε το θέμα των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη και αλλού βέβαια, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, ακόμα ταυτοποιήσει τα του της ε, και επιβάλλει πολύ δαπανηρές ε, δομές σε ρυθμιστικό επίπεδο, πράγμα το οποίο επιβαρύνει την ανταγωνιστική κότητα μάλλον του τομέα. Επίσης, όταν μιλάμε για πρόσβαση της αγοράς σε, με χώρες Ασεάν ή του περσικού κόλπου, είναι σαφές ότι θα έπρεπε να υπάρχει αμοιβαιότητα της πρόσβασης. Αυτό είναι τμήμα της απελευθέρωσης. Και εδώ έρχομαι και στο θέμα του κ. Ερτούγκ. Τι θα κάνουμε με τις χώρες του ΑΣΕΑΝ ή του Περσικού κόλπου. Θέλουμε απλά και μόνο διαφάνεια και αμοιβαιότητα πρόσβαση στην αγορά, ένα θεμητό ανταγωνισμό. Αυτές είναι βασικές ε, και θεμελιώδεις αρχές. Και τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Όσον αφορά τους κανόνες του ανταγωνισμού, έχουμε καλό παραδείγματα από την Κομισιόν και τα κάτι μέλη που χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες στις συναλλαγές με τα κράτη εκτός Ένωσης. Ε, είναι πολύ ευέλικτο αυτό το ε, πλάνο και η Κομισιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτά που, στοιχεία που θεωρεί ότι είναι τα πιο κατάλληλα για αυτήν την συγκεκριμένη επαφή και σχέση. Πιστεύω πως η διαφάνεια, ανεξαρτητή έλεγχη, είναι δύο από τους βασικούς ε, παράγοντες κλειδιά. Φυσικά θα πρέπει πάντα να κοιτάμε την πρόσβαση στην αγορά και τέτοια πράγματα, αλλά όταν μιλάμε για διατήρηση της ακυριότητας της ευρωπαϊκής ιστορικής αγοράς και περί αυτού είναι ο λόγος σήμερα, θα έλεγα ότι πάντοτε η, ε, η διαφάνεια και η ανεξάρτητη έλεγχη είναι τα βασικότερα. Σε σχέση με τις εναλλακτικέ απόψεις της αεροπλοείας, υπάρχουν πολλά που κάνει η βιομηχανία της αεροπλοείας και έχει ήδη κάνει. Ε, Ε, παίρνει πολύ καιρό το να εξασφαλιστούν εναλλακτικά καύσιμα τα οποία να είναι ασφαλή και εδώ θα έχουμε πολύ ε, μεγάλο όφελες. Οι ευρωπαϊκές ε, αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν 10 με 20 δις το χρόνο σε φόρους. Φανταστείτε αν μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να επανεπενδύσουμε στα προϊόντα μας και στην βιωσιμότητα του τομέα. Ε, πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα. Και αυτό βέβαια και σε σχέση με τις παρατηρήσεις της κυρίας Ντέλη. Ε, αυτά από μένα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ο, ο κύριος Τζον Χάνλον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαντενκάμπ. Όχι, δεν έχουμε καταρχήν ε, συμμαζέψει το σπίτι μας. Έχουμε πιστεύω τεράστιο δυναμικό σε εμπορικό εταίρο στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς ε, ο κατακαιρματισμός ε, και η διχόνια μεταξύ μας ε, αξιοποιείται από τους άλλους παγκοσμίους εταίρους μας. Τώρα, για τις κρατικές ενισχύσεις υποτιθέμενες. Και εμείς στην Ευρώπη έχουμε κρατικές ενισχύσεις ή ήδη κρατικών ενισχύσεων ε, ενίσχυση κρατικών ε. αερογραμμών, ε, επιδοτούμενα δάνεια και εταιρείε που δεν είναι βιώσιμες και παρα, παρόλα αυτά παραμένουν στην αγορά. Τέτοιου είδους φαινόμενα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και δεν έχουν τη θέση τους σε μια πραγματικά ελεύθερη αγορά. Το θέμα των κρατικών ενισχύσεων δεν συνδέεται μόνο με τις εταιρείε χαμηλού κόστους γιατί ακούμε ότι δίνονται κρατικέ ενισχύσει σε περιφερειακά αεροδρόμια. Οι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναθεωρηθεί και μα ικανοποιούν οι νέε, γιατί υπογραμμίζουν την ανάγκη να υιοθετηθεί η οικονομία τη αγορά και αρχέ ε, για τι επενδύσει στην οικονομία τη αγορά. Και θα πρέπει ε, οι αεροδρομικές, οι αεροπορικές εταιρείες να λειτουργούν ως ε, συνετοί επενδυτές και δεν έχουμε προβλήματα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το θέμα έχει αντιμετωπιστεί και η έκβαση των συζητήσεων μας ικανοποίησε. Για το περιβάλλον, μόνο εμείς ήμασταν υπέρ ενός μηχανισμού της αγοράς και το ευρωπαϊκό ETS ήταν αρχικά καλό. Αν όμως θέλουμε να συνεχίσουμε, ε, να δώσουμε, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες άδειες, αλλιώς θα τις αγοράσει κανείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός είναι καλός, αλλά η συρρήκνωση του πεδίου εφαρμογή τη τον κατέστησαν αναποτελεσματικό. Και παρεκτράπημεν από την πορεία μας αρχικά και από τον πραγματικό σκοπό του ETS. Τώρα όλοι περιμένουν καλύτερη έκβαση των διαπραγματεύσεων στο ΙΚΑΟ. Ελπίζω να ευοδοθούν. Αλλιώς πραγματικά θα σκάψουμε μόνοι μας το λάκκο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις προσπάθειές μας για τα καύσιμα. Και είναι ενδιαφέρον ότι εστιαζόμαστε στις αεροπορικές εταιρείε όταν μιλούμε για τα καύσιμα. Γιατί όμως ε, δεν ε, μιλούμε και για τις δικές μας εταιρείε και για τις, ε, τα υπέρογκα κονδύλια που δίνονται στην έρευνα. Γιατί μόνο ένα καύσιμο έχουμε για την αεροπορία, την κυροζίνη. τη χρησιμοποιούμε όσο πιο ορθολογικά γίνεται και παρόλα αυτά μας τιμωρούν για τις εκπομπές μας. Ενώ μια πετρελαϊκή εταιρεία ξοδεύει τεράστια κονδύλια για την έρευνα και ε, αξιοποιεί τα αποτελέσματα, ενώ εμείς μόνο ένα καύσιμο έχουμε και δεν έχουμε δυνατότητα για ε, αλλαγή. Ο κύριος Πόλοτσεκ. Ευχαριστώ. Έρχομαι στο ερώτημα του κύριου Φάντερ Κάμπ. Η KLM με έδρα το Άμστερνταμ έχει φτιάξει μια νέα συμφωνία <clears throat> με τους ε, ε, πιλότους μείωσε το συνολικό κόστος του πιλωτηρίου κατά 15%. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε σωστές λύσεις μαζί με τους εργαζομένους σε ένα ανοιχτό κοινωνικό διάλογο. Αλλά ο κοινωνικός διάλογος όταν έχουμε πιλότους οι οποίοι εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ενώ αν δεν είναι οι πιλότους που βρίσκονται σε πουλ όταν τους λέμε θα πρέπει να είστε πιο πιο φτηνή κτλ. Εκεί δεν συμφωνούμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται καθόλου όταν είναι άρρωστοι. Όταν είναι χωρίς ε, δουλειά δεν έχουν καμία κάλυψη καθόλου. Έχουν μαϊμού θέσεις, έδρες πολλές φορές για να μειώσουν τις ε, συνεισφορές του κοινωνικού τομέα. Αυτή είναι η μαύρη πλευρά λοιπόν, η σκοτεινή πλευρά της κατάστασης και το pay to fly, το σύστημα αυτό που πληρώνει κανείς για να μπορεί να βρίσκεται σε μια θέση στο πιλωτήριο για να μπορέσουν να μπουν στην, ε, στον τομέα αυτό Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Αυτό είναι τμήμα του αθέμητου ανταγωνισμού. Στο ερώτημα της Γκεζίνε Μάιστερ, <coughs> πώς να εξασφαλίσουμε την ισότητα ανταγωνισμού. Αυτό το κέριο ερώτημα, δώσατε τμήματα, ψήγματα της απάντησης. Θα πρέπει να έχουμε σωστές Μιλάτε όχι μόνο για το με τον αεροπορικό τομέα, αλλά και για τους κατασκευαστές των αεροσκαφών. Και αυτό είναι τμήμα του προβλήματος. Πουλάει πάρα πολλά αεροπλάνα η έρμπα στον πεσικό κόλπο. Δεν έχει κανένα συμφέρον να υπάρξει ισότητα ανταγωνισμού. Πολλές φορές λέμε ότι η έρμπα εξαρτάται από αυτή την αγορά. Η Emirates έχει 140 α380 σε παραγγελίες, 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ χοντρά λεφτά. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε μια κοινωνική ρήτρα στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών. Με την πρώτη ευκαιρία αυτή η παράγραφος δεν πέρασε την πραγματική δοκιμασία. Γιατί μια νορβηγική εταιρεία έδωσε έδρα στους πιλότους της και το πλήρωμα καμπίνας στην Μπανκόκ που φυσικά ήταν μια μαϊμού βάση για να αποφύγουν το υψηλό φορολογικό και κοινωνικό κόστος στην ε, Νορβηγία. Οι ταϊλανδικές αρχές δεν είχαν ιδέα για όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο εμεί βασιστήκαμε στην παράφο 15 στη Συμφωνία Ανοιχτών Εθέρων Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και δεν λειτουργήσε από ευρωπαϊκή πλευρά. οι αμερικανικέ εταιρείε, η αμερικανική δικαιοσύνη είπε όχι σε αυτό το πράγμα. Είπε ακριβώς γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η παράγραφος. Αν εμεί θεωρούμε ότι δεν είναι στεναρή η θέση μα για τον τομέα αυτό που φέρνει πολλά ωφέλη σε επίπεδο ΑΕΠ, σε επίπεδο εισοδήματο των Ευρωπαίων, εάν εμεί. δεν, δεν εκμεταλλευόμαστε και δεν αξιολογούμε σωστά αυτό, τότε έχουμε λάθος στις προτεραιότητες μας για μένα. Ο καθένας εδώ εκπροσωπεί τον εαυτό του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μερικά κοινά σημεία. Παραγματικά για τους ανοιχτούς ευρωπαϊκούς εθέρες. Αυτό είναι κάτι που να προχωρήσει. Είπατε για τη Φραγκφούρτη. Σας ενόχλησε που η Φραγκφούρτη έχει υποσκελιστεί από την Κωνσταντινούπολη. Έξι ώρες την ημέρα, το 24ωρο, είναι κλειστό το αεροδρόμιο της ε, Φραγκφούρτης και πριν από αυτές τις 6 ώρες υπάρχουν περιορισμοί πτήσεων. Έχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο σενάριο που έχει βοηθήσει τις χώρες του Περσικού κόλπου και τις τουρκικές αερογραμμές. Ναι, ναι, σύντομα θα τελειώσω. Δεν υπάρχει λοιπόν σε κανένα σημείο ισότητα ανταγωνισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολιβιέ Γιάνκοβιτς σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, οι ερωτήσεις ήταν ε, πολύ ε, θετικές. Θα θέλαμε να δούμε όντως ανοιχτή πρόσβαση στις αγορές, να δούμε την απελευθέρωση της ιδιοκτησίας και τον έλεγχο των εταιριών σε αμοιβαία βάση. Αυτά όλα θα έχουν την τυποποίηση της βιομηχανίας της και πιστεύω πως το θεμελιώδες θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με την έννοια ότι δεν θα μπορέσουμε όπως η Ευρώπη, στην Ευρώπη να επιβάλλουμε στον υπόλοιπο κόσμο τους δικούς μας εσωτερικούς κανόνες ιδιαίτερα όταν τμήμα αυτών των εσωτερικών κανόνων δημιουργούν ε, μειον, ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε ολόκληρο τον τομέα της αεροπλοείας. Αυτό που είναι σημαντικό, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, ε, είναι να ταυτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Ε, και εδώ μπορεί να κάνει πολλά κομισιόν, αλλά όταν δεν κάνει σε λεπτομέρειες όλα αυτά τα ζητήματα, θεωρώ πως πολλά εξαρτώνται από το εθνικό επίπεδο, από τα κράτη-μέλη. Πώς λοιπόν θα κατευθύνουμε τα κράτη-μέλη ώστε να ε, ενεργήσουν προς την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Και έπειτα, κρατικές ενισχύσεις. Εγώ θα εστιάσω ιδιαίτερα στο θέμα της δημόσιας χρηματοδότησης των υποδομών. Πριν από 10 χρόνια η Κομισιόν θεωρούσε πως η δημόσια χρηματοδότηση στις υποδομές των αεροδρομίων αποτελούσε ένα μέτρο οικονομικής πολιτικής και ότι δεν ε, σήμαινε κρατική ενίσχυση. Τώρα έχουμε αλλάξει τη θέση μας. Τώρα Όντως οι υποδομές οι αεροπορικές μπορούν να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση, αλλά είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν μαζικές δημόσιες επενδύσεις στις αεροπορικές υποδομές ε, και αυτό φυσικά ε, δεν βοηθά να είναι πιο ανταγωνιστικό ο τομέα. Να δούμε την τιμολόγηση μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων, όπω ανέφερε και ο Τζον. Ξέρετε, αν δεν μπορείς ε, να χρηματοδοτήσεις ε, δημόσια, το τίμημα της χρήσης των υποδομών θα είναι και μεγαλύτερο. Το ίδιο και για την ασφάλεια. Πάλι στην Ευρώπη εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν χρηματοδοτούμε δημόσια την ασφάλεια της αεροπορίας. Τα αεροδρόμια μετατρέπονται σε τεράστιες εταιρείες ασφάλειας. Πριν από την 9η ε, Σεπτεμβρίου στο, ε, ήμασταν στο 5% ε, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στο 20% λειτουργικό κόστος το οποίο παροφά η ασφάλεια. Τα άλλα αεροδρόμια δεν έχουν αυτό το κόστος, άρα και οι τιμές τους δεν είναι τόσο ψηλές. Πολλή δουλειά λοιπόν πρέπει να γίνει και ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τους ίδιους μας τους κανονισμούς. Τέλος για να κλείσω, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ε, η αγορά κινείται. Ο κόσμος ε, κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με αυτές τις εντολές που ζητά η Κομισιόν. Συζητάμε για το ποια προτεραιότητα θα πρέπει να θεσπίσουμε. Εγώ νομίζω πως όλες οι εντολές αυτές είναι προτεραιότητα και αυτό επίσης ε, θίγει το θέμα των πόρων εντός της Κομισιόν για το πώς δηλαδή θα μπορέσει η Κομισιόν να χειριστεί το θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κλάους Γκάιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω στον κύριο Έρτουγκ για την ερώτηση ποιο τμήμα είναι σημαντικό στην πραγματεύση με την ΑΣΕΑΝ. Η ΑΣΕΑΝ είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά με πληθυσμό 600 εκατομμύρια ανθρώπους και μάλιστα προσπαθεί να αναπτύξει μια ενιαία αεροπορική αγορά, κάτι που έχουμε κάνει και εμείς στην Ευρώπη, οπότε μπορούμε να έχουμε τέτοιου του συμφωνία, block to block όπως λέμε. Και οι άμεσες ροές επιβατών μεταξύ Ευρώπης και Ασεάν ήταν σταθερή τα τελευταία χρόνια, αλλά η πραγματική κυκλοφορία έχει αυξηθεί ετησίως κατά 5% την τελευταία δεκαετία. Όλη αυτή όμως η αύξηση ε, πέρασε από κόμβους ε, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής. Δεν πέρασε από ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οπότε θέλουμε πραγματική εταιρική σχέση με την περιοχή ΑΣΕΑΝ για να ενισχύσουμε τις απευθείας ε, συνδέσεις και να ανακτήσουμε μερίδια αγορά που έχασαν οι αεροπορικέ μα εταιρείε. Την τελευταία διετία είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ΑΣΕΑΝ. Συγκρίναμε τι πολιτικές μας σε θέματα αεροπορία και ε, ανακαλύψαμε πολλά κοινά σημεία στου στόχους, στι πολιτικές και του στόχους των πολιτικών μα. Είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν ότι η ΑΣΕΑΝ θα ενδιαφερθεί και ήδη έχει ξεκινήσει μια κανονιστική ευθυγράμμιση. Πιστεύουμε ότι θα υλοποιήσουμε τις αρχές του θεμητού ανταγωνισμού. Έχουμε κάποια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ πάντως θα στηρίξει την ανάπτυξή μας και στην ΑΣΕΑΝ. Και μεταφορά εμπορευμάτων ε, έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό προσπαθούμε να, επιδιω... υλοποιήσουμε τη συμφωνία για να βελτιώσουμε και τη μεταφορά εμπορευμάτων, την αεροπορική. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Μάισνερ για τον ΙΚΑΟ, ε, εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μαζί με τα κράτη-μέλη το έργο της ΚΑΟ προκειμένου να θεσπιστεί ένα πολυμερές πλαίσιο για την ε, απελευθέρωση του διακτησιακού καθεστώτος ε, και την εφαρμογή των αρχών της αγοράς ε, και τον έλεγχο των αεροπορικών εταιριών. Πάντως είναι μια πολυσχηδής διαδικασία και θα είναι και χρονοβόρα. Θα εφηγραμμιστεί μάλλον προς τα κάτω Πάντως πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει να εξαγάγει τα κανονιστικά της πρότυπα και τις προδιαγραφές και στα θέματα της αεροπορίας. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Νταλή, για το περιβάλλον, ε, πιστεύω ότι η, διάσκεψη, η διάσκεψη των Παρισίων δημιούργησε μία όθηση θετική και άσκησε πίεση σε ολόκληρο τον κλάδο. Η αεροπορία με μια συνεκτική προσέγγιση που έχει η τεχνολογία για τα καύσιμα κάνει, έχει σημειώσει πρόοδο και η πρόταση για τους νέους ευρωπαϊκούς εθέρες θα συμβάλλει τα μάλα και ως προς την πτυχή αυτή. Τώρα έχουμε το 2016 τη διάσκεψη της ΙΚΑΟ. Δεν θα θέλαμε να αποτύχει αυτή, γιατί αν ξαναποτύχει η ΙΚΑΟ θα δημιουργηθεί αβεβαιότητα, κάτι που ε, δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Αν μας μείνει χρόνος αργότερα θα αναπτύξω κάποια κοινωνικά θέματα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών, 22 ε, μήνες πέρασαν και περιμένουμε άδειε με βάση την κοινοτική νομοθεσία το θέμα της, είναι θέμα ακαιρεότητας της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη περιμένουμε εξηγήσει από την ΆΗ. Και προσπαθούμε να εγγύψουμε στα κοινωνικά θέματα, αλλά θα επανέλθω σε αυτά αργότερα, αν μείνει χρόνος. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ακόμα από τα μέλη της Επιτροπής. Ο Γκάλε ο Γιαούτο, Κλούν, η Ίνες Αγιάρα Σέντερ. Now, Isabel de Monte und ich. Fast alle, Όλοι δηλαδή οι παρόντε περίπου. Ενάμιση λεπτό ο καθένας, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι για να υπάρχει χρόνος για την απάντηση. Ο Μικαέλ Γκάλεν, ο πρώτος ευχαριστώ, είναι τόσο πολλά τα οποία έχουν λεχθεί. Θα μιλήσω συνθηματικά και τηλεγραφικά. Η NEA εθέρες. Εδώ τα εμπόδια βρίσκονται από, στα, από την πλευρά των κρατών μελών που θέλουν να προστατεύσουν ορισμένα συνδικάτα πολλές φορές. Εσείς μπορείτε να ασκήσετε πίεση στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν οι NEA εθέρες για λόγους ασφάλειας, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για λόγους ασφάλειας ακόμα. Επίσης για τα, τους φραγμούς η Κομισιόν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. αλλά δεν αφορά μονάχα τις ε, ιδιωτικές εταιρείε, αλλά και τα κράτη-μέλη. Εσείς έχετε κάνει κάτι για τη χώρα μου σε ό,τι αφορά το φόρο ε, για τις ε, αεροπορικές εταιρείε. Και ένα τρίτο ερώτημα, ένα θέμα το οποίο δεν τίθεται καθόλου όταν μιλάμε για την ισότητα ανταγωνισμού. Βλέπετε κάπου κάποιος από εσάς τη δυνατότητα οι κανόνες του ΠΟΕ να εφαρμοστούν και στον αεροπορικό κλάδο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολιτικά επιθυμητό, είναι κάτι που το θέλει η Κομισιόν. Γιατί αν δεν μπορέσουν να εφαρμοστούν οι κανόνες του ΠΟΕ, τουλάχιστον να ενσωματώσουμε κάποιους από αυτούς τους κανόνες στις διμερείς συμφωνίες για να μπορέσουμε σταδιακά να οδηγήσουμε σε ανοιχτούς εθέρες. Ευχαριστώ και ιδίως γιατί ήταν σύντομος. Τα παντέλου. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. πριν από την συνάντηση αυτή είχαμε ήδη σκεφτεί πως υπάρχει το πρόβλημα των αεροπορικών εταιριών των χωρών του Περσικού Κόλπου, ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε για θέμη τον ανταγωνισμό ε, και το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω αυτών των εταιριών. Πολλές ε, διαδρομές που καλύπτονταν παλιότερα από ευρωπαϊκές εταιρείε τώρα έχουν ε, καταληφθεί από τις εταιρείε του Περσικού και αυτό είναι δικό προς δικό τους όφελος γιατί είναι ελληνικές εταιρείε ε, οι οποίες χαίρουν επιδοτήσεων, κρατικών ενισχύσεων, ε, έχουν επιδοτήσεις, ε, έχουν πρόσβαση στις υποδομές, στο κεφάλαιο και στα καύσιμα με μεγάλη ευκολία. Πιστεύετε πως το πακέτο που παρουσιάστηκε στις 16 Δεκεμβρίου ασχολείται αποτελεσματικά με την απώλεια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών γιατί είναι εύκολο να πείτε όχι ή ναι, αλλά ε, συμπληρωματικά θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του νομοθετικού πακέτου προς αυτή την κατεύθυνση και ως χρήστης των διαφόρων υπηρεσιών. Μιλήσαμε για ανταγωνιστικότητα, για ωφέλη τα οποία έχουν ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες. Μιλήσαμε για θέσεις απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τους επιβάτες και τα δικαιώματα αυτών. Σκεφτείτε το και αυτό, διότι αυτές οι εταιρείες ε,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 θόλης της ύλη, από τον κύριο Πόλατσεκ που δεν θέλει να δει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε ξένα χέρια, ε, στον κύριο ε, Γκάιλ, που μίλησε για συνολικές καθολικές συμφωνίες. Ε, εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Νομίζω όμως ότι εκτός από τον κύριο Γιάνκοβιτς όλοι μιλήσατε είτε για ίσους όρους του παιχνιδιού, είτε είναι αυτό παραπλανητικό είτε όχι, πάντως όλοι ε, αναφέρθηκατε σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ε, εντάξει, κανείς δεν θα διαφωνήσει μαζί σας. Μόνο όμως ο κύριος Γιάνκοβιτς μας δίνει κάπως ε, μια πιο στρατηγική εικόνα και απάντησε και τις ερωτήσεις μας πιο λεπτομερώς. για το ποιο είναι ο αθέμητο ανταγωνισμό από αυτέ τι εταιρείε, Τι εκμεταλλεύονται δηλαδή ακριβώ που δεν μπορούν να το κάνουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε στην ευρωπαϊκή αγορά. λαμβάνοντα υπόψη ότι ορισμένε από αυτέ τι εταιρείε ε, χαίρουν κρατικών ενισχύσεων. Όλοι θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό, σαφώ να το ταυτοποιήσουμε τα του οίκου μα. Αλλά τι έχουν αυτοί παραπάνω που εμεί δεν έχουμε στην ευρωπαϊκή αγορά. Danke Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ένα κομμάτι της ερώτησής μου ήδη καλύφθηκε από τους συναδέλφους, αυτό που σχετίζεται με τις κρατικές ενισχύσει και προσπάθησα να κάνω την ίδια ερώτηση στην Επίτροπο Πούλτς πριν από λίγες μέρες αλλά δεν πήρα απάντηση. Αναμένοντας ο ΙΚΑΟ να υιοθετήσει διεθνείς κανόνες για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή για τις μαζικές χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ευρω... από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ε, στις ευρωπαϊκές εταιρείες άλλων εταιριών που ε, παίρνουν μεγάλες κρατικέ ενισχύσει στις χώρες τους. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει, δεν υιοθετεί νόμους για να προστατέψει τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την υπόθεση του χαμηλού κόστους. Εδώ γενικότερα θα πρέπει να συζητήσουμε την, πλοήγηση, την, την αεροπλοεία ως μέσο μεταφοράς. Γίνεται κερδοφορία και κερδοσκοπία στην πλάτη των πολιτών. Πώς γίνεται το ίδιο ταξίδι να κοστίζει 50 ευρώ και σε μια, για μια άλλη 1000 ευρώ. Ε, από τη μια πλευρά είναι εξαιρετικά χαμηλά η τιμή με προβλήματα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε αυτή την εταιρεία, την ασφάλεια κτλ. Και από την άλλη έχουμε μια τιμή που είναι προφανώς εξαιρετικά υψηλή και άρα ε, κερδοσκοπεί πάνω στην πλάτη των ε, επιβατών, των πελατών εντάξει ανταγωνισμός, αλλά για ορισμένου τομεί, με ορισμένε περιοχές, όπως οι νησιωτικές ας πούμε, ή ειδικά από απομακρυσμένες, θα πρέπει να θεωρηθεί και, εντάξει, όχι η δημόσια υπηρεσία, αλλά εν γιατί πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας μεγαλύτερος έλεγχος όσον αφορά τη συνοχή των τιμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο Λούν. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν και την ε, σαφή παρουσίαση των θέσεών τους. Πολλές απορίες μου ήδη απαντήθηκαν. Μίλησαμε για θεμετό ανταγωνισμό. Είναι καλύτερος και πιο δόκιμος όρος από τον ισότιμο ανταγωνισμό, γιατί η ισότιμη ανταγωνισμού είναι ουτοπία. Οι επενδύσεις έχουν γίνει από αεροπορικέ εταιρείε και όπω έδειξε ο χάρτη τον κύριο Ιακωβέτση είδαμε ποιοι νέοι ε, δρόμοι ανοίγουν, ποια νέα δρομολόγια. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε λοιπόν γιατί ο κόσμο είναι μικρό με την παγκοσμιοποίηση. Η συνδεσιμότητα λοιπόν αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για όλους και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες. Η αεροπορική συνδεσιμότητα θα έχει ζωτική σημασία και κέριο ρόλο. Επίσης, ε, είναι κρίμα που δεν εντάσσεται και οι αεροπορία συμφωνίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού 868, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι θα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση το 2016, αλλά φοβάστε μήπως καθυστερήσει λόγω της ε, καθυστέρησης άλλων συμφωνιών στον ίδιο τομέα. Επίσης μίλησατε πολύ θετικά για το δυναμικό της επικείμενης συμφωνίας με την ΑΣΕΑΝ λόγω των κοινών μας σημείων. Υπάρχουν άλλες περιοχές του κόσμου με τις οποίες σχεδιάζεται, με τις οποίες σχεδιάζεται παρόμοιες συμφωνίες. Περσικός κόλπος για παράδειγμα, η Τουρκία. Γιατί είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη και τα αεροδρόμια τους λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Δεν κλείνουν καθόλου όπως τα δικά μας, οπότε από εκεί ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Πού βλέπετε άλλες δυνητικές συμφωνίες που θα μας δώσουν ευκαιρίες και πρόοδο στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ινές Αγιάλα Σέντα. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές και να τους ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας θέσανε και να, και να θέσω κάποια ερωτήματα. Μιλάμε για τον αθέμητο ανταγωνισμό των εταιριών του Περσικού Κόλπου. Όχι μόνο των εταιριών αλλά και των αεροδρομίων. μέσα σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς <clears throat> είναι να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, συμφωνίες και τις συνθήκες μας. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, σίγουρα έχουν μια τέτοια στεναρή αντιμετώπιση, προστατεύουν τις αξίες τους όπου είναι αυτό ε, απαραίτητο. Δεν είναι κατά ανάγκη κακός ο προστατευτισμός όταν προασπίζει τις αξίες μας στα κοινωνικά θέματα, στο περιβάλλον, στα θέματα ισότητας δεν υπάρχει μονάχα κακός προστατευτισμός. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι και να αφήσουμε τις χώρες αυτές και τις εταιρείε να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο που δεν δέχονται την ανοιχτή αγορά. Θέλω όμως εσείς να μας πείτε από την Κομισιόν ή από την και εσείς και η Κομισιόν αν πραγματικά είναι τελείως ανέφικτο να υπάρξει η ισότητα ανταγωνισμού. Εμείς έχουμε πάντα την ε, θέληση να έχουμε ίσες ε, ευκαιρίες για όλους στον υγεία, στην παιδεία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει το βασικό πλαίσιο στις διεθνείς συμφωνίες να είναι η ισότητα ευκαιριών. Αλλιώς πάμε σπίτια μας. Δεν μπορεί να λέει τώρα η ε, <clears throat> Επιτροπή ότι είναι όλοι διαφορετικοί όπως τα δάχτυλα του χεριού που λέγανε πάλι. Εντάξει, αλλά να, τουλάχιστον να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Αλλιώς θα γίνει αυτό που είναι και με ε, δραστηριότητες όπως η Φαντουργία που τα βγάλαμε τελείως από την Ευρώπη και τώρα οι Ισπανοί εργάζονται ως ε, έχουν φύγει από την δραστηριότητα αυτή και δουλεύουν μονάχα άνθρωποι ως σκλάβοι για να παραγάγουν υφάσματα. Παρακαλώ εσείς που έχετε μια ευθύνη, κάντε κάτι ναι, το καταλάβαμε, λέει ο πρόεδρος. Μην μακρηγορείτε άλλο. Η κυρία Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας για αυτά που είπανε. Και πολλά έχουν ελεχθεί ήδη από πολλά λύσαντες. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα την ε, αξιολόγησή σας για το, λόγο, το, ρόλο που μπορεί να παίξει η διεθνής, ο διεθνής ανταγωνισμός για το πακέτο αυτό το αεροπορικό που προτείνει η Κομισιόν που θα πρέπει να μας εξασφαλίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ασφάλεια. Και επίσης για τις ε, εταιρείε κατασκευαστικού χαρακτήρα να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά των ευρωπαϊκών εταιρών. Αυτό σημαίνει <clears throat> να έχουν και περισσότερη ε, φιλελευθερωποίηση των ε, κατασκευαστικών του εταιριών. Πού μπορεί να δοθεί η έμφαση εδώ. Ευχαριστώ. Φυσικά πολλές ε, παρατηρήσεις έγιναν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορίας που σχετίζεται και με τις ικανότητες, την ικανότητα των Ευρωπαίων να δράσουμε ε, για τα δικαιώματα των επιβατών, για τα τέλη αεροπορίου, αεροδρομίου, για την συμφόρηση, για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. Έχουμε βέβαια ακόμη όμως κάποια κρεμή προβλήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω έκκληση και στους Ισπανούς συναδέλφους μετά τις Ισπανικές εκλογές να το λάβουν αυτό υπόψη και να συμβάλλουν και αυτοί στην ανέβρεση λύσης και να ασκήσουν πιέσεις. Όχι αν είχαμε και κανένα Βρετανό συνάδελφο στην αίθουσα, θα πέφτει έκκληση και στους Βρετανούς. Να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε λύσεις και να μείνουμε ενωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Δεύτερη παρέτηση. Τώρα θα αφήσουμε το θέμα, δεν θα ανοίξω το θέμα του Γιβραλτάρ. Επίσης, θα πρέπει να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες, να εντείνουμε τις προσπάθειες για σφαιρικές συμφωνίες με έξυπνο τρόπο, να αναζητήσουμε παγκόσμιου μηχανισμούς. Προτιμώ να δουλεύαμε στο πλαίσιο του ΠΟΕ για παγκόσμιου μηχανισμούς και όχι μόνο στον ΙΚΑΟ. Και τέλος, σημαντικό όμω, η αναθεώρηση του κανονισμού 868. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει κάποια αποτελέσματα και χαίρομαι που το υποσχέθηκε για το Μάρτιο. Βλέπω μια υποσημείωση στο έγγραφο Στρατηγική που αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει υπό τον όρο του ευνομοθετήν. Η νομοθεσία να αναθεωρηθεί εφόσον είναι καλύτερη. Οπότε ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει έργο και να το κάνει το συντομότερο δυνατό αποφεύγοντας ε, τον μπλοκάρισμα και τον κύριο Τίμερμαν. Γιατί θα πρέπει και τον 868 να συζητήσουμε. Ιζαμπέλ Ντεμόντε ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και να παρατηρήσω την αλήθεια ότι υπάρχουν ε, τέλη αεροπορικά τέλη, αλλά πολύ συχνά αυτά χρησιμοποιούνται και ως κίνητρο για να έχει κανεί συγκεκριμένες διαδρομές. Ε, στον κύριο Χάνλο όμως θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ε, σε σχέση με το όσο είπε ο κ. Πολούτσι για την κατάσταση των πιλότων. Να πω να ρωτήσω ποια είναι η διάσταση του φαινομένου που αφορά ορισμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται όπως ας πούμε το pay to fly όπως εδώ ήδη έγινε μνήμα σε αυτό, αλλά και στα προσωρινά συμβόλαια, αλλά και συμβάσεις μηδενικών ορών, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν ε, εταιρείε που ε, έχουν φορολογική έδρα σε ένα κράτος μέλος, ενώ έχουν βάση έδρα αλλού, πραγματική έδρα αλλού. Και αυτό βεβαίως για να ευνοηθούν από το φορολογικό καθεστώς της εν λόγω χώρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσας ακρόαση. Θα προσπαθήσω να παραμείνω σε επίπεδο ρεαλιστικό. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα σε όλους για το θέμα της εφαρμογής της τωρινή οδηγίας. Το ερώτημα μου το εξή: Αν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, κάτι που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη, αν δημιουργήσουμε του ενιαίου εθέρε που αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένοι και τα κράτη-μέλη δεν κάνουν καμία προσπάθεια να ξεπεράσουν αυτόν τον κατακαιρματισμό. Πόσα από τα προβλήματα που έχουμε ενώπιό μα θα μπορούσαμε να επιλύσουμε, γιατί μιλάμε πολλά για τη θέση κομισιών, για τη ρύθμιση, για την αναθεώρηση. Τι γίνεται αν δεν εφαρμοστούν όμω όλα αυτά. Τι κάνουμε εμεί με τα κράτη-μέλη. Του ζητάμε να τηρήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για να μειώσουν τον κατακαιρματισμό και να ξεπεράσουμε το ένα δισεκατομμύριο που χάνουμε σε καινοτομία λόγω αυτού του κατακαιρματισμού γιατί ένα μεγάλο μέρος της αεροφυγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την καινοτομία. Για μένα είναι ένας τομέας ο οποίος είναι στρατηγικός. Εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά, όχι μονάχα η αναγωνιστικότητα αλλά και ο ρόλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το ερώτημα μου είναι απλό λοιπόν. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα αυτό τι ζητάτε από τα κράτη-μέλη. <clears throat> Του ζητάμε να τηρήσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν το κάνουν. Του ζητάμε να κάνουν του ενιαίου εθέρε. Δεν το κάνουν. Είμαστε μόνοι τελικά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι από τα πρώτα θέματα που πρέπει να επιλύσουμε. Αφορά και τον αεροπορικό κλάδο και σε άλλου τομεί. Δεν είμαστε πιο ανταγωνιστικοί γιατί δεν θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και θα ήθελα μια αξιολόγηση από εσά γιατί αυτό με απασχολεί. Πώς μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες με διαφάνεια όταν εμείς από μόνοι μας αποθούμε τη διαφάνεια. Μιλάμε για συμφωνίες με τρίτες χώρες και ρήτρες που πρέπει να τεθούν και νιώθουμε άγχος γιατί δεν μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά αλλά δεν επιλύουμε τα θέματα που αφορούν το εσωτερικό μας. Μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι που δεν είναι ρεαλιστικό, πρέπει να είμαστε πιο τίμοι, πιο ρεαλιστικοί και να θέσουμε τα ερωτήματα πραγματικά σε εσωτερικό επίπεδο. Ιδίως αν θέλουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό τομέα και θέσεις εργασίας ποιότητας και μια διάσταση του αεροπορικού κλάδου που να αξίζει να την αξίζουν οι πολίτες μας. Ευχαριστώ και εγώ ζήτησα να λάβω το λόγο. και έχω ακούσει για τις επιδοτήσεις προς τις ε, αεροπορικές εταιρείες μέσω της μη πληρωμής ΦΠΑ και της ε, αφορολόγητης κυροζήνης. Αυτό μονάχα εξηγείται ότι έχουμε 3.000 πτήσεις κάθε χρόνο μεταξύ Στουτγάρδης και Φραγκφούρτης που δεν είναι μεγάλη απόσταση. Έχουμε την ε, συνεδρίαση για το κλίμα που λέει ότι πρέπει να μειώσουμε τις πτήσεις και να λύσουμε προβλήματα στα αεροδρόμια. Όχι με περισσότερες πτήσεις, με λιγότερες πτήσεις και όχι με πτήσεις που δεν τις χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και το ερώτημά μου. Αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο πρέπει να αφορά το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι <clears throat> έχουμε και καλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ τρόπων μεταφορών. Δεύτερο, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες οι ευρωπαϊκές εταιρείε δεν μπορούν να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως τα καταφέρουν τα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Αυτό λοιπόν είναι ένα ήδη καλό, κακό παράδειγμα γιατί αν δεν μπορούμε να τα βρούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουμε να τα βρούμε και με τα κράτη του πεσκού ε, κόλπου. Και επίσης θα ήθελα <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι οι ανοιχτοί εθέρες ισχύουν και στις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά μας να συμμετάσχουν όλες αυτές οι χώρες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Και τελευταίο ερώτημα. Γιατί ξαφνικά στα εταιρείε χαμηλού κόστους συμμετέχει η British Airways εκεί και όχι η Lufthansa ή η Air France. Δεν καταλαβαίνω γιατί η British Airways έχει προνομιακή σχέση με τις εταιρείε χαμηλού κόστους. Και πάλι με την ίδια σειρά σας δίνω την ευκαιρία να απαντήσετε. Δύο λεπτά θα σας δώσω τώρα στον καθένα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα τις ερωτήσεις για την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Φαίνεται ότι οι χώρες μέλη του ΠΟΕ δεν θέλουν να συμπεριληφθεί η αεροπορία στις συμφωνίες του ΠΟΕ. Μόνο τρεις ίσορες σημασίες πτυχές των υπηρεσιών έβαλαν μέσα. Επίσης, ε, ε, τα, οι καταναλωτές ε, έχουν δείξει προτιμήσεις τους και αυτό κάνουν σε μια ανοιχτή αγορά. Για τα κέρδη. Όταν μιλούμε για θέμητο ανταγωνισμού θα πρέπει να επιλαμβάνονται οι εθνικές αρχές και για την αθέμητη τιμολογιακή πολιτική για παράδειγμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική θέση, την πολιτική τους, ε, με την πρόθεση των κόμμων τους. Είπατε λιγότερη αεροπορία. Η δική τους πολιτική είναι περισσότερη αεροπορία, περισσότερες πτήσεις. Και επίσης έχουν πολύ καλύτερες βάσεις, σε πολύ χαμηλότερο κόστος και από αυτή την άποψη έχουν πολύ μεγαλύτερο όφελος. Τώρα, για την διαφανή τιμολόγηση. Ε, δύο ευρώ την πτήση χρεώνουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι αν έχουμε μια ανοιχτή πολιτική τιμών θα έχουμε και νέους ερχόμενους που θα προσφέρουν νέα προϊόντα και άρα μεγαλύτερη επιλογή στον καταναλωτή. Αυτό είναι το όφελος μιας ανοιχτής αγοράς. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός φιλόσοφος Νάκη, ε, μιλάτε για τους Ευρωπαίους, ε, νέους ευρωπαϊκούς εθέρες. Κάντε το επιτέλους, αφήστε τα λόγια. Πρέπει να περάσουμε στα έργα, να προχωρήσουμε πέρασε η ώρα, 10 δευτερόλεπτα μου, έλειψα, μου έμειναν. Μιλήσατε για την ισότιμο ανταγωνισμό και είπατε είναι ευκαιρία. Μια πραγματικά θεωρητική ε, όμως κατάσταση είναι και αν δεν έχουμε ποιοτικέ υπηρεσίες δεν θα υλοποιηθεί. Όλοι οι αεροπορικές εταιρείε θα πρέπει να έχουν στην ίδια αγορά τις ίδιες ευκαιρίες. Έχουμε όμως νικητές και ιτημένους. Δεν είναι θέμα μεριδιού αγορά, αλλά ικανότητα ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Καλύφθηκε το θέμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Κυρία Ταπαρδέλ, ε, αν είναι αρκετό το πακέτο, όχι με την παρούσα μορφή. Αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σημασία του κλάδου. Ωραία, είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, το στηρίζουμε, αλλά να φανεί αυτό συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσο προχωρά το πακέτο. Ε, δεν αρκεί ακόμη, ελπίζουμε στο μέλλον να ολοκληρωθεί. Κύριε Τελίτσκα, για τα κέρδη. Είναι ένα συνδυασμό μια στρατηγική πολιτική προσέγγιση για το τι εστί αεροπορία και ποια είναι η προστιθέμενη τη αξία στην κοινωνία. Αυτό λείπει στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όχι τουλάχιστον στο μέτρο που το βλέπουμε σε άλλε χώρε, σε άλλου εταίρου. Ε, πολλοί ομιλητέ περιορίστηκαν στι χώρε του κόλπου, αλλά έχουμε και άλλα καλά παραδείγματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, όταν βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν τις υποδομές, ε, ε, τα αεροδρόμια ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, οπότε έχουν την ευκαιρία για μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών τους στα αεροδρόμια. Ενώ στην, ε, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λειτουργούν 16 με 17 ώρες τη μέρα πώς να μην υπάρχει πίωση της αγοράς ε, και πώς θα κάνουν βιώσιμες τις εργασίες τους. Επίσης, ε, κυκλοφορούν συνέχεια φήμες για την ε, επιβολή φόρου στα καύσιμα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, ούτε θα εμπλακώ σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλά ανησυχητικά θέματα εκεί. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Τώρα, εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Πολλά παραδείγματα έχουμε εδώ, το μίλησαν και οι συνάδελφοι, Ευρωπαίοι, ενιαίοι ευρωπαϊκοί εθέρες, συγγνώμη, να εφαρμοστεί η πρόταση. Έχουμε πολύ καλά περιβαλλοντικά μέτρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν. Και τέλος, κύριε Κράμερ, ευχαρίστως να έχουμε τη συζήτηση για την αεροπορία και τις ενισχύσεις, κρατικές ενισχύσεις, ε, φορολογία στα καύσιμα. Πολύ ωραία να γίνει συζήτηση, αλλά να λάβουμε υπόψη όλα τα μέσα μεταφοράς και όλες τις πτυχές, ε, τις υποδομές, τον ηλεκτρισμό, την ενέργεια, τους φόρους. Μιλούμε για ε, ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων μεταφοράς, αλλά αν γίνει συζήτηση, να είναι σφαιρική και να καλύψει και όλες τις πτυχέ και όλα τα μέσα μεταφοράς. Πάντως, καλό θα ήταν να γίνει στο μέλλον. Ο κύριο Χάνλον. Ευχαριστώ. Τι έχουν αυτοί που εμείς δεν έχουμε. Ε, προσωπική μου άποψη, αν και μπορεί να είναι επίμαχη, έχουμε ένα παρελθόν. Έχουμε τη δυνατότητα ε, να κυριαρχήσουμε την αγορά λόγω έλλειψης ανταγωνισμού από την άλλη ε, πλευρά της διαδρομής. Διμερείς συμφωνίες που δεν τις απελευθερώσαμε ήταν εκεί ε, για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τις αγορές. Γι' αυτό ακριβώς και στηρίζουμε τόσο πολύ το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι συνθήκες ε, στις οποίες λειτουργούν έχουν σπάσει την αγορά, έχουν εφεύρει, έχουν και ενοτομήσει, έχουν διαρκώς την προσοχή τους στο ε, τι θέλει ο πελάτης. Δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να μορμουράμε. Καλύτερα είναι να μάθουμε από αυτό. Αν έχουμε πρόβλημα με την ιστορία μας και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα, όχι το δικό τους. Έπειτα, για... Εγώ είμαι αρκετά ανήσυχο όταν ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξάγει τις ρυθμιστικές της αρχές σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το προσπαθήσαμε αυτό με το ETS και δυστυχώς κολλήσαμε. Ε, αυτή τη δικασία λοιπόν έχει ξεκινήσει σε επίπεδο του ΙΚΑΟ. Υπάρχουν ομάδες εργασίας για ε, το ρυθμιστικό πάνελ. Θα είναι πραγωγικό νομίζω αν υπάρχουν κάποιες παγκόσμιες προδιαγραφές, αλλά όχι περιφερειακή λύση δεν νομίζω πως αυτή είναι η πραγματική απάντηση και πάνω απ' όλα δεν θα πρέπει αυτή η διαδικασία να φρενάρει το να συνεχίσουμε τις, τις, την απελευθέρωση συμφωνιών ή την σύναψη συμφωνιών. Ίσως ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι η ΚΑΟ θα έχει αυτό το ρόλο να καθυστερήσει τη διαδικασία και να περιορίσει τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποια ερώτηση. Αν το έκανα, σας ζητώ συγγνώμη των προτέρων. Για την British Airways ε, δεν είπατε τίποτα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το θέμα, δεν κατάλαβα. Σας έθεσε το ερώτημα για την British Airways. Η British Airways είναι τώρα εταιρεία χαμηλού κόστους. <coughs> ναι. Καλώς ήλθανε. Εμείς αν ε, ζητήσουν να έρθουν, δεν θα τους λέγαμε όχι. Η British Airways παρουσιάζει τον εαυτό τους πελάτες της ως εταιρεία χαμηλού κόστους. Η Vueling είναι μέλος μας για τρία χρόνια και συμμεριστεί τις αρχές μας, αλλά πιστεύουν στον ελεύθερο ανταγωνισμό και έχουν 119 πτήσεις το, τη, μέρα, τη βδομάδα από το Μπρεσικό κόλπο στην ε, Αγγλία δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, ενώ η Γαλλία που έχει 32 μόνο τέτοιες πτήσεις διαμαρτύρεται τα, ε, τα μάλλον. Κύριος Πόλατσακ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που ξέχασα άνοιξω το μικρόφωνο για τις ε, πτυχές που έχουν να κάνουν την αναθεώρηση του 868 και τις διαπραγματεύσεις. Η ρήτρα θεμητού ανταγωνισμού που βρίσκεται στην, ε, στο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας είναι ένα σημαντικό βήμα σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ανοιχτών εθέρων ή αεροπορικού χαρακτήρα συμφωνίες, ότι πετυχαίνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Και πάλι νομίζω λοιπόν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θέση ισχύω και όχι αδυναμίας, γιατί η πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε σημαντικη κυριε για τον κατάλογο των αθέμητων πλέον εκτιμάτων έναντι της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού κλάδου από την πλευρά των ΗΠΑ. Από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο οποίο εμείς να έχουμε ένα πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε φτηνή εργασία, σε φτηνή χρηματοδότηση. για να χρηματοδοτηθούν αγορές από την Airbus, της χάρη. Και η δική μας γεωγραφική θέση δεν είναι ευνοϊκή. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα για αυτά τα θέματα, προς το παρόν τουλάχιστον. Η κυρία Ιούτο αναφέρθηκε στις ε, οι γεωγραφικές θέσεις κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Στην Κύπρο η Ερσάιπρος, η πρώην εθνική εταιρεία, χρεοκόπησε. Και η Μάλευ στην Ουγγαρία χρεοκόπησε. Εμείς είδαμε τι έγινε με το εθνικό εισόδημα και ζητήσαμε από τους αδέρφους μας στην Κύπρο να κάνουν το ίδιο. Κοιτάξτε τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στο ΑΕΠ να δείτε αν υπάρχει κάποια επίπτωση. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας το είχαμε δει αυτό. Μετά από την ε, χρεοκοπία της ε, Μάλευ μειώθηκε κατά 3% το εθνικό εισόδημα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του αεροπορικού κλάδου. Ένα καλό παράδειγμα στο ερώτημα της κυρίας Μπιλμπάου για τον έλεγχο και την ιδιοκτησία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Όπως ξέρετε, τα δικαιώματα πτήσης είναι διμερεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Περσικού κόλπου. Αλλά για να έχει κάνει τα δικαιώματα πτήσης, για να τα περιορίσει μάλλον, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν. Για την Air Berlin στη Γερμανία υπήρχαν κάποιες διαδρομές που δεν καλυπτόντουσαν από δικαιώματα πτήσης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Και τώρα ο Ολιβιέ Γιάνκοβιτς. Ευχαριστώ. Για το θέμα τι έχουν οι χώρες του Περσικού κόλπου που δεν το έχουμε εμείς. Μα γεωγραφική θέση, πολύ σημαντική. Νομίζω αυτό τους δίνει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και ε, για χρόνια ολόκληρα δεν το αξιοποιούσαν. Τώρα το αξιοποιούν και δημιουργούν και μόχλευση. Υπάρχει και το θέμα βέβαια των κρατικών ενισχύσεων, επενδύσει στις υποδομές, την ασφάλεια, το είπα και προηγουμένως. Μόνο με τους δικούς μας κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και με την επιβολή τους προς τα έξω δεν θα το πετύχουμε. Γιατί τα δημόσια κονδύλια στις επενδύσεις στις υποδομές και οι δημόσιες επενδύσεις των μέτρων ασφάλειας είναι θεμητά εργαλεία, αλλά δημιουργούν ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ένα στοιχείο από το 2012. Στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το κόστος ε, της ασφάλειας της αεροπορίας ήταν 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Τα στοιχεία των αεροπορικών εταιριών σε ό,τι αφορά τα άμεσα τέλη που έδιναν ήταν 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η δημόσια ενίσχυση της ασφάλειας ε, ως ανταγωνιστικού παράγοντος. Τώρα, έχουμε διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και μεγάλο κατακαιρματισμό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σε μια συνολική συμφωνία για την αεροπορία. Είναι τμήμα της οικονομικής πολιτικής και των στόχων. Ε, και λογικό να μην το έχουμε. Τώρα, τι στερούνται εκείνοι που το έχουμε εμείς. Ε, εμείς έχουμε τέλη και φόρους της, ε, τη φορολογία της αεροπορίας που μας ταλανίζουν. Συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Αυτό που φταίει με τις συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού είναι ότι είναι παραπλανητικό αυτό το θέμα και δεν μας ε, οδηγεί εκεί που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι ο θεμητός ανταγωνισμός. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, μιλήστε για την ανάγκη περιορισμού των πτήσεων δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της αεροπορίας για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική της θέση και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Και είμαστε όλο και περισσότερο εξαρτημένοι από το εξωτερικό εμπόριο. Και αν θέλουμε να στέλνουμε τα προϊόντα μας στον Νέα στο Johannesburg ή αλλού, δεν θα τα στείλουμε σιδηροδρομικός, αλλά αεροπορικός εννοείται. Επίσης, ε, ενισχύσεις ε, στα άλλα μέσα μεταφοράς. Θέλουμε ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Και σίγουρα ο σιδηροδρομικός κράτος παίρνει 42 δισεκατομμύρια ενισχύσεις. Ε, είναι υπέρογο το ποσό. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μειωθεί για να έχουμε ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων μεταφοράς. Ο κύριος Γκάιλ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις διατυπώθηκαν. Θα ξεκινήσω από αυτές της κυρίας Κλούν. Ρωτήσατε, κυρία Κλούν, αν η πρόταση για την αναθεώρηση του 868... Α, έφυγε η ενδιαφερόμενη. Αν θα καθυστερήσει την πρόοδο ε, της χορήγησης εντολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εντολών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι η αναθεώρηση του 868 είναι δικαιολογημένη και η χορήγηση εντολής ε, θα μπορούσε να καθυστερήσει αντίθετα αν δεν υποβάλαμε πρόταση αναθεώρηση το 868. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι κάποιες χώρες και κάποιοι ε, συντελεστές της αγοράς ε, ανησυχούν τα μάλα για τις αθέμετες πρακτικές. Και αυτό που θέλουμε στην συνολική συμφωνία είναι να μην επικεντρωθούμε μόνο στις χώρες του κόλπου, γιατί πολλές ε, προτάσεις ε, δεν αφορούν συγκεκριμένες χώρες, είναι μέσα και μηχανισμοί που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να θωρακιστεί απέναντι στις αθέμητες εμπορικέ πρακτικές οποιασδήποτε χώρας του κόσμου. Και θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της παροχής δικλείδων ασφαλείας για να αποσοβήσουμε τις αμφιβολίες και ε, να αντισκεδάσουμε τους φόβους κάποιων, ε, ιδιαίτερα χωρών μελών που παγάωσαν το, τη χορήγηση δικαιωμάτων πτήσεων και να ενισχύσουμε περαιτέρω την, ε, το άνοιγμα των αγορών που είναι υπέρ των καταναλωτών. Με ταυτόχρονα όμως μέτρα υπέρ της ασφάλειας. Είχαμε επικοδομητικό διάλογο και με την ΑΣΕΑΝ, όπως είπα, και βρήκαμε κοινά σημεία. αυτό θα επιδιώξουμε και στη συναντήσεις μας και συμφωνίες με την Τουρκία και τις χώρες του κόλπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη και ελκυστική ε, αγορά. Σε αυτή διεισδύουν πολλές αεροπορικές εταιρείες και τους ενδιαφέρει να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο. Και φυσικά δεν θα πρέπει να γίνει ανεφόρον αυτή η εισαγωγή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει να τηρούν τους όρους. Η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη χώρα. Ε, μεγάλη επίσης χώρα με μεγάλη ε, και ταχαίως αναπτυσσόμενη αεροπορία και έχουμε ξεκινήσει στήρη συνεργασία με τη χώρα αυτή και νομίζω ότι και οι χώρες του Περσικού κόλπου έχουν τέτοια συμφέροντα και ενδιαφέρον για περαιτέρω συμφωνία. Τώρα, ο ρόλος της ΕΑΣΑ στο διεθνή ανταγωνισμό. Η στρατηγική μας για την αεροπορία τάσεται υπέρ μια, ενός ισχυρού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας με ισχυρό ρόλο και διεθνώς και τη χρησιμοποιούμε σε όλα τα προγράμματα παροχής τεχνογνωσία στον κόσμο. Και επίσης προτείνουμε αναθεώρηση του βασικού κανονισμού της ΕΑΣΑ, προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της με απότερο σκοπό, ε, γιατί όχι και για μια ενιαία ευρωπαϊκής αρχής πολιτικής αεροπορίας. Αυτά και αν έχετε περισσότερες απορίες μπορούμε να βρεθούμε και εκτός της συνεδρίασης. Πολλά σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Είχαμε σκεφτεί ότι ίσως ήταν πρόβλημα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση τόσο κοντά στα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά ήταν επιτυχής, ήταν ιδιαίτερα εμπλουτιστικέ οι παρουσιάσεις και σας ε, εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και να ευχηθώ στους βουλευτές, ε, τους ε, συνεργάτες και θα έχουμε ένα μικρό ποτό μετά. Είσαστε όλοι καλεσμένοι. Καλά Χριστούγεννα και ευχαριστώ.